Πάλι καλά κατάφερα και πάτσα το σωστό κουμπί τόσα χρόνια που είμαι εδώ. Καλώ ήρθατε λοιπόν στη συνεδρίαση τη Επιτροπή, ε, τη Επιτροπή Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων. Αν δεν έχετε παρατηρήσει, μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Δεν βλέπω παρατηρήσει. Ούτε αντιρρήσει για την ημερήσια διάταξη και αν δεν υπάρχουν και για τα πρακτικά, τότε τα έχουμε εγκρίνει έω το τέλο τη συνεδρίασή μα. Και ενημερώνω ότι θα υπάρξει μετάδοση μέσω του διαδικτύου της συνεδρίασης με το σύστημα του web streaming. Έχουμε ανακοινώσει γραμματείας για την έκτακτη συνεδρίαση της 22 της, ημέρα, της 22 ε, Νοεμβρίου για ανταλλαγή απόψεων ως προς την έκθεση της κυρίας Ρόιτεν ε, για τις συντάξεις έχουν επίσης ενημερωθεί οι συνάδελφοι για την παράταση συνεδρία τη Δευτέρα Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, από τι 3 έω 6.30. Επίση, θα δείτε το έγγραφο 11, του 2010 ω προ τα θέματα του, των μη των ε, παρατηρητών ή των ειδικών μάλλον χωρίς δικαίωμα ψήφου για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κατάρτισης που έχει την Γραμματεία. Επίσης θα δείτε από τη Γραμματεία μας ερώτηση προς την Επιτροπή για τις εφαρμογές του EGF και θα δείτε σε ποιες χώρες αναφέρεται. Το πρώτο θέμα που έχουμε στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση της ε, κυρίας Τσίμερ για την φτώχεια των γυναικών και ύστερα από την συνεδρίαση που είχαμε την προηγούμενη φορά και την ε, ένσταση επί του διαδικαστικού ορισμένων συναδέλφων, έγινε συνάντηση μεταξύ συγγητηρία και σκιωδών συγγητών, όπου συμφωνήθηκε το ορισμένο και των ε, τροπολογιών που είχαν κρυθεί έτσι με τον ε, κανονισμό, θα γίνουν αποδεκτές. Γνωρίζω δε ότι είμαι, είναι ενήμεροι και οι συγγήτρια αλλά και οι σκιώδεις συγγητές για το ποιες είναι αυτές οι τροπολογίες. Αυτά ως προς τις ανακοινώσεις μου και παρακαλώ την Καμπρίελα Τσίμερ να κάνει την ε, παρουσίαση της εκθεσής της και των τροπολογιών. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, ευχαριστώ τους συναδέλφους της Επιτροπής μας που συνέπραξαν σε αυτή τη γνωμοδότηση και που έδειξαν και την ε, καλή διάθεση να ξαναδιαπραγματευθούν μαζί μου τα όσα μπορούσαμε να θεωρήσουμε αποδεκτά, παραδεκτά καλύτερα ή μη στην έκθεση αυτή και πράγματα τα οποία μπορούν να, και, να βρουν και σύμφωνα την Επιτροπή των Γυναικών. Ιδιαίτερα σε ευχαριστώ πολύ και την Πρόεδρο της Επιτροπής των Γυναικών η οποία εξασφάλισε το να έχουμε μια ε, καταγραφή όχι υποκειμενική αλλά αντικειμενική των ε, προτάσεων που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω ότι όλες οι τροπολογίες για τις οποίες ε, εξέφρασαν τη συμφωνία οι συντάκτες τους κατατίθενται σαν μια γενική δήλωση της Επιτροπής μας ή μια ανακοίνωση, αν θέλετε, κατά της φτώχειας των γυναικών ανά τον κόσμο ως πρόταση προς την Επιτροπή των Γυναικών. Υπάρχει και ένα μικρό κόλπο, θα έλεγα, ότι δηλαδή σε ορισμένες περιπτώσεις προσδιορίζουμε ότι πληττόμενοι από τη φτώχεια είναι εν προκειμένου όχι αποκλειστικά, όχι εν τη ευρία έννοια οι γυναίκες, αλλά οι πιο ηλικιωμένες, οι πιο ηλικιωμένοι και εδώ ευχαριστώ ιδιαίτερως τα μέλη της Επιτροπής. Εν γέννη, με βάση τις που έγιναν αποδεκτές, που κρίθηκαν παραδεκτές και με τους σκιώδεις συγκητές, καταλήξαμε να διαπραγματευτούμε μία σειρά πέντε συμβαστικών τροπολογιών και πάλι ευχαριστώ ιδιαίτερω για τη συνεργασία. Συμβαστικές λοιπόν τροπολογίες οι οποίες ε, κατ' είναι απλές, χωρίς προστριβές δηλαδή τροπολογίες, γιατί εκφράζουν την πλειονότητα των κατατεθισών τροπολογιών. Και έτσι μπόρεσαν να εμπνεύσουν τις ε, ε, συμβαστικές τροπολογίες να ενταχθούν σε αυτές. Τις έχετε λοιπόν τις συμβαστικές αυτές τροπολογίες. Φαντάζομαι στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας ε, τις ε, λάβατε. Δύο ιδιαιτέρως παρουσιάζουν κάποιες ανακρίβειες ή σφάλματα ίσως θα έλεγα. Στη συμβαστική τροπολογία υπαριθμών Β, παραδείγματι, είχαμε ακόμα σήμερα το πρωί ε, διαπραγματεύσει μεταξύ δύο βουλευτών, την κυρία Λόπε Φοντάνα και την κυρία Ιώτοβα συγκεκριμένα, οι οποίες θα επεδίωκαν ε, συμβιβαστική πρόταση. Από την κυρία Ιώτοβα έχω μία απάντηση, αλλά από την κυρία Λόπα Φοντάνια δεν έχω επίσημη ε, επιβεβαίωση ότι έχετε συμφωνήσει και γι' αυτό έχω προσωρινά περιλάβει στον κατάλογο των ε, συμβαστικών τροπολογιών αυτή την πρόταση, περιμένοντας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης την επιβεβαίωση ε, ότι είναι αποδεκτή. Εδώ μιλούμε για την συμπερίληψη του όρου ή μάλλον της διατύπωσης ε, σε αποτελεσματική χρήση και επίσης του όρου κοινωνικής προστασίας αντικοινωνικής ενσωμάτωσης. Δεν έχω αντίρρηση ως προς τις παρατηρήσεις αυτές. Απλώς θα ήταν σημαντικό και πάλι να είμαστε βέβαιοι ότι ε, καλύπτονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι από την διατύπωση αυτή. Και γι' αυτό περιμένω από το γραφείο της κυρίας Φοντάνη την επιβεβαίωση ότι όντως ε, συνήθει αυτή η συμφωνία, ότι υπάρχει αυτή η συνεργατική λύση. Για την Α, Γ και Δ, C και D δηλαδή, την περιλαμβάνουμε όπως ακριβώς είχαν διατυπώσει το κείμενο οι συντακτές, συντακτρίες καλύτερα, για τη συμβαστική ε θα ήθελα να σημειώσω ότι λυπούμε ιδιαίτερο το λέω ρητά αυτό, διότι κατατέθηκε αυτή η πρόταση και εδώ έχουμε να κάνουμε μια συμβαστική η οποία ασχολείται, πραγματεύεται καλύτερα την μελέτη που είχε κατατεθεί στην Επιτροπή μας, την ε, κοινωνική προστασία ως σταθεροποιητή σε συγκυρία, σε δεδομένη συγκυρία, συγκυριακό μάλλον σταθεροποιείται Έχετε υπόψη σε αυτή την έκθεση. Πλην όμως δεν την έχουμε λάβει όλοι γραπτός και ως εκ τούτου θα ήθελα να αποφύγουμε σε τέτοια περίπτωση και στην γνωμοδότηση αυτή φράσεις οι οποίες ενδεχομένως να δημιουργούν προβλήματα. Δηλαδή λέγεται ότι μπορεί να έχουν μεγαλύτερο ε, σταθεροποιητικό ρόλο από τις ε, κλασικές κυβερνητικές ή κρατικές δαπάνες αυτά τα μέτρα. Έτσι είναι αυτή η φράση και παραλαμβάνω δεν θέλω να έχω πρόβλημα στη συνέχεια γιατί θα διαπιστώσω ότι κάτι διαφορετικό προκύπτει από αυτή τη μελέτη. Παρακαλώ τους αδέλφους να δείξουν κατανόηση. Γενικά η πρόταση νομίζω δεν είναι κακή αλλά θα ήθελα να διαγραφεί σε αυτό το σημείο και σε αυτή την έκδοση του κειμένου. Και άλλωστε στο κείμενο που σα έστειλα λίγο πριν τις 3 το έχω αναφέρει, απλώς δεν ξέρω αν το έχετε λάβει. Για την ε, εξέλιξη των διαπραγματεύσεων τώρα. Βλέπω ότι συμφωνούν οι περισσότεροι με τις συμβαστικές τροπολογίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την υποστήριξη αυτή και να σημειώσω ότι έχουμε να κάνουμε από εδώ και μπρος μια σειρά ε, διευκρινήσεων, καλύτερων διατυπώσεων, προκειμένου να βελτιωθεί το κείμενο. Έχουμε μια σειρά άλλων ε, τροπολογιών τώρα, οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί από τις συμβαστικές, τις οποίες συνιστώ να εγκρίνουμε πλην εκείνων ε, τις οποίες δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω δεκτές, της κυρίας Γκέρλινγκ, και δεν μπορούσα να περιλάβω και στις συμβαστικές, διότι βρίσκονται σε αντίθεση, ευθεία αντίθεση με τα όσα έχω εγώ προσπαθήσει να κάνω ως συντάκτρια και μέσα από τις συμβαστικές τροπολογίες. Θα ήταν δηλαδή αντιφατικά με τα υπόλοιπα του σχεδίου γνωμοδότης, με τα υπόλοιπα κομμάτια του σχεδίου γνωμοδότης, αλλά και με τις συμβαστικές τροπολογίες. Βλέπω ότι η κυρία Γκέρινγκ από την ECR έχει τελείως διαφορετική άποψη για, τα, για τις θέσεις που εκφράζω εγώ και γι' αυτό δεν μπορώ να τις συμπεριλάβω στις συμβαστικέ μου τροπολογίες. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Όπως είπα, ήταν ουσιαστικά δύο οι τροπολογίες τις οποίες χρειάζεται να γίνει μια μικρή μετατροπή. Και για τη Β, όπως είπα, περιμένω την οριστική επιβεβαίωση από την κυρία Λόπε Φοντάνια ότι έχει συμφωνήσει. Ευχαριστούμε. Η κυρία Νίλσον και η κυρία Λόπες. Η κυρία Νίλσον. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα να θίξω δύο ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, συμφωνώ απολύτως με την εισηγήτρια για την τροπολογία 42, για τους δείκτες, για την ένδια. Και εγώ η ίδια Έχω υποβάλει μια τροπολογία σχετικά. Διότι αυτό που κυρίως με ανησυχεί είναι ότι τα κράτη-μέλη θα κάνουν κατάχρηση της ελευθερίας τους. Χρησιμοποιώντας τρία διαφορετικά σύνολα δεκτών ταυτόχρονα. Προκειμένου να μην κάνουν όλα όσα προβλέπεται να κάνουν για να καταπολεμήσουν την ένδια και για να, ωραίο, να καλοποιήσουν μάλλον τα αριθμητικά του στοιχεία. Είναι πιο εύκολο να καταπολεμάται έτσι η φτώχεια παρά να ασχολείται κανεί με του ανθρώπου που βγαίνουν εκτό αγορά εργασία ή είναι θύματα τη δομική ένδυα. Εδώ λοιπόν στηρίζω την εισηγήτρια. Για την συμβεβαστική Β, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Υπάρχουν κάποια καλά στοιχεία εδώ, όμως έχουμε πρόβλημα ιδίω με τη μνήα της αύξησης στην χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. αυτό είναι δύσκολο να το στηρίξουμε, έτσι όπως αναφέρεται, και ελπίζαμε ότι θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε κατά τμήματα εδώ. Θα αποφασίσουμε. Νομίζουμε ότι είναι ένα τελείως άλλο θέμα αυτό. Θα πρέπει να το δούμε στην ομάδα εργασίας CGF. Τα συζητάμε και αυτά. Συζητάμε και την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση που θα γίνει του χρόνου. Και νομίζω ότι θα ήταν για μας σε μια τόσο σημαντική έκθεση να έχουμε αυτή την μνήμα. Α μην το αναφέρουμε ίσως. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λόπε Φοντανιέ. Εμείς θα θέλαμε καταρχάς να συγχαρούμε την ε, εισηγήτρια, γιατί νομίζω ότι όλες οι πολιτικές ομάδες συνεργάστηκαν πολύ καλά. Καταλήξαμε σε συμφωνία και το σχέδιο έκθεσης που θα παρουσιαστεί μου φαίνεται πολύ καλύτερο από αυτό που θα περιμέναμε αρχικά. Σε σχέση τώρα με τις συμβιβαστικέ τροπολογίες, σε σχέση με την Β, την B Βεβαίως, ε, διαπραγματευτήκαμε, ζητήσαμε κοινωνική ένταξη αντί για κοινωνική προστασία, γιατί το κοινωνική προστασία κατά τη γνώμη μας δημιουργούσε ένα πρόβλημα επικουρικότητας και άκουσα την εισηγήτρια και την ευχαριστώ για αυτά που είπε σχετικά. Τώρα, μετά από την τροποποίηση αυτή, εμείς υπερψηφίσαμε την, ε, υπερψηφίζουμε αυτήν την συμβιβαστική τροπολογία. Τώρα, εμείς είμαστε υπέρ της αύξησης ε, του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε σε περίπτωση που μας την αρνηθούν. Όσον αφορά τη συμβιβαστική τροπολογία ή e, θα καταψηφίσουμε, σας το λέμε από τώρα. Γιατί δεν πιστεύουμε ότι η κοινωνική προστασία είναι ένας σταθεροποιητής είτε των εσόδων είτε των εξόδων. Άκουσα όμως την εισηγήτρια που μόλις μας είπε ότι θα αποσύρει την παράγραφο αυτή, οπότε εμείς αν αποσυρθεί η παράγραφο αυτή, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Μπορούμε να υπερψηφίσουμε το υπόλοιπο τη συμβιβαστική τροπολογία ή. Αυτά ήθελα να πω. Και να σα υπενθυμίσω μόνο ότι εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν σε μία έκθεση για την ε, φτώχεια των γυναικών, αρνούμαστε να χρησιμοποιήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη γυναίκα. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Στάινερ. Η κυρία Ιώτοβα, που δεν μπορούσε να έρθει σήμερα, με παρακάλεσε να την εκπροσωπήσω για να διατυπώσω τα σχόλιά της. Μου τα έτοιμασε στα αγγλικά και γι' αυτό επιτρέψτε μου να σας διαβάσω το αγγλικό κείμενο. Θα ήθελε η κυρία Γιώτοβα καταρχά να ευχαριστήσει την, την συντάκτρια και του κύριους συγητέ ε, για την προετοιμασία τη εκθέση τη χρηματοδοτήσεως. Η κυρία Γιώτοβα είναι εν γέννη ικανοποιημένη με τι τροπολογίε και τι συμβαστικέ τροπολογίε. Φρονεί ότι έχουμε μπορέσει να ενσωματώσουμε όλε τι δύσκολε πτυχέ και τα σημαντικά σημεία στι ε, τροπολογίε, έτσι ώστε να συμβάλλουμε στη διατύπωση μια καλή έκθεση, γνωμοδότηση μάλλον ε, για την έκθεση της Επιτροπής των Γυναικών, της κατουσίαν αρμόδιας ε, Επιτροπής, έτσι ώστε να ε, θέσουμε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τη φτώχεια των γυναικών και τον αγώνα για την απαλλαγή από τη φτώχεια. Η κυρία Ιώτοβα πιστεύει ότι η κατάλληλη ενίσχυση της χρηματοδότησης ε, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού ε, ταμείου για την Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση των δύο ταμείων είναι απαραίτητη προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση για τους φτωχότερους και εκείνους που κινδυνεύουν, για τους φτωχούς και εκείνους που κινδυνεύουν να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας ε, και γενικά σε όσους ζουν σε συνθήκες αβεβαιότητας ένα ζήτημα σχετικό με τις αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ένωση προ την παροχή κοινωνική προστασία που έχει τεθεί. Υποχρεώνει την κυρία Ιώτοβα να καταθέσει μια προφορική τροπολογία η οποία αντικαθιστά την κοινωνική προστασία με την κοινωνική ενσωμάτωση προκειμένου να, αποτραπεί ο κίνδυνος ε, παρερμηνίας ε, ή προβλήματα επικουρικότητας. Κατά τα άλλα, με τις ε, προτάσεις και τις συμβαστικές τροπολογίες δεν έχει προβλήματα η κυρία Ιώτοβα. Ευχαριστώ η κυρία Γκρίνερ, λοιπόν, και κυρία... πρώτα όμως η κυρία Μοραντζάτ. Μογά Σαχτιέ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς ε, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Τσίμερ, αλλά να ευχαριστήσω και τους σχεώδες εισηγητές κυρία την, κυρίως την ε, σκιώδη συγγήτρια κυρία Λοπές Φοντανιέ, γιατί για το θέμα αυτών των τροπολογιών, ε, για την έκθεση αυτή, κάναμε πολύ σημαντική δουλειά. Μου φαινόταν βέβαια λίγο παράξενη όλη η διαδικασία, γιατί όλες οι τροπολογίες τη επιτροπή Απασχόλησης δεν θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνουν ε, τον όρο γυναίκα, γιατί μόνο η Επιτροπή Γυναικών μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτόν τον όρο στις τροπολογίες της. Αν είχαμε παραμείνει εκεί, θα φτάναμε στο παράλογο και μάλιστα πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους, όλους όσους συμμετείχαν σε αυτήν ε, την ε, ε, παράξενη συνάντηση. Μπορέσαμε με ευφυή τρόπο να εξασφαλίσουμε όλες οι τροπολογίες ε, της Επιτροπής Απασχόλησης ε, να μπορούν πραγματικά να παρουσιαστούν εκ μέρους της Επιτροπής Απασχόλησης και να είναι και ουσιαστικές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν τους συμμετέχοντες και κυρίως γιατί είναι πραγματικά και ένα μάθημα για το μέλλον ε, σε σχέση με τις εργασίες μας και σε σχέση με τις εργασίες της Επιτροπής Γυναικών. Και όταν βέβαια ε, μιλάμε για την φτώχεια των γυναικών, νομίζω ότι μπορούμε να επικεντρωθούμε και στα θέματα της απασχόλησης. Είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό. Υποβάλαμε πολλές τροπολογίες, ε, η Πασκάλ Γκρινή ε, και εγώ συνεργαστήκαμε πολύ καλά. Θα πάρει και εκείνη το λόγο άλλωστε να μας πει περισσότερο για το θέμα αυτό, γιατί όλο μιλούσαμε για την κοινωνική βοήθεια, για την κοινωνική προστασία, για όλα αυτά τα θέματα και αυτό που είναι σημαντικό είναι να αναγνωρίσουμε σήμερα ότι η φτώχεια των γυναικών προέρχεται αυτή τη στιγμή από την επαγγελματική ένταξη, την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Δηλαδή, αυτό είναι ο βασικό λόγο τη φτώχεια του, αυτό είναι ο βασικό παράγοντα και έχουμε λοιπόν έναν αριθμό τροπολογιών που υποστηρίζουν ακριβώς αυτήν την επαγγελματική ένταξη ούτως πίν, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την κοινωνική ένταξη. Η κοινωνική ένταξη είναι μία συνέπεια της ένταξης των γυναικών από επαγγελματικής απόψης και είναι κάτι που για μας είναι εξαιρετικά σημαντικό. Στις τροπολογίες Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι διαφορές ε, αμοιβή ανδρών και γυναικών ε, θα μειωθούν. Είναι και αυτό ένα τμήμα της, ε, του αγώνα κατά της φτώχειας των γυναικών. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό στοιχείο στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε και πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί ώστε τα προγράμματα κατάρτισης διαβίου εκμάθησης να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά και μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση, γιατί μεταξύ της επαγγελματική του ζωής, της οικογένειακή του ζωής και της διαβίου εκμάθησης και λόγω όλων αυτών μπορεί να υπάρξουν ε, διακρίσει και πάλι ει βάρο των γυναικών. Οπότε θα ήθελα να επενθυμίσω σε όλους ότι οι τροπολογίες που δεν υποβάλλονται ε, στην εκ μέρους της Επιτροπής ε, Απασχόλησης θα υποβληθούν στην Επιτροπή Γυναικών. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκρουνή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω ε, και την εισηγήτρια την κυρία Τσίμερ αλλά και ε, όλους τους κοιόπους εισηγητές και την συνάδελφο Βερόνικα, ε, την Βερόνικα Λόπε Φοντανιέ, η οποία μας υποστήριξε πάρα πολύ για τη συμβιβαστική τροπολογία B. Εγώ συμφωνώ με τη διαγραφή της κοινωνικής προστασίας, άλλωστε νομίζω ότι μας το επιβεβαίωσε και την ευχαριστούμε. Όσον αφορά τώρα το... Ε, ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο. Όλο και περισσότερα ζητούμε συνεχώς ε, για να λάβουμε λιγότερα όμως, ε, γιατί πρόκειται για ένα στοιχείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συμφωνώ λοιπόν απολύτως ε, με την συνάδελφο Ελισαβέτ Μορέν Σαρτιέ, γιατί δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν να χρειαστεί να, να τροποποιήσουμε τις δικές μας τροπολογίες για να μην χρησιμοποιούμε την λέξη γυναίκα από τη στιγμή που ούτως ή άλλως ο σκηνός μας στόχος είναι το να μην υπάρχει πια η γυναική αυτόχεια. Και δεν καταλαβαίνω επίσης πώς είναι δυνατόν να μην γίνεται αποδεκτή τροπολογία μου υπαριθμών 54 που αφορά ε, τις απολύσεις για τις γυναίκες, ε, Δηλαδή να, είναι να δοθεί προτεραιότητα στις γυναίκες οι οποίες έχουν ε, ακριβώς μεγάλα οικογενειακά βάρη και δεν είναι δυνατόν λοιπόν αν χρησιμοποιούμε τον όρο απασχόληση πρέπει να μπορούμε να χρησιμοποιούμε και τον όρο γυναίκα. Διαφορετικά δεν υπάρχει κανένα νόημα να υποβληθεί η τροπολογία αυτή. Εν πάση περιπτώσει η τροπολογία υπαριθμό 54 εντάξει θα υποβληθεί στην Επιτροπή Γυναικών αλλά βρίσκω ότι είναι κρίμα πραγματικά γιατί είναι δική μας αρμοδιότητα το θέμα αυτό της απασχόλησης των γυναικών. Και ευχαριστώ πάρα πολύ ε, τους γιατί όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, τα σημεία που με απασχολούσαν, τελικά βρήκαν τη θέση τους τροπολογίες. Τέλος, λέει η Πρόεδρος, η κυρία Χάρκιν, πριν ε, ε, δώσω το λόγο και πάλι στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Η κυρία Μάιντσνερ ε, θα μας πει περισσότερα, γιατί μόλις ήρθε και θέλει να κάνει μερικά σχόλια. ναι, να δώσουμε το λόγο στην κυρία Μάισνερ και μετά η κυρία Γκρουνέρ. Ε, ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Στο συγγνώμη που ήρθα με τόση καθυστέρηση. Έχω τρει ταυτόχρονε συνεδριάσει σήμερα. Είναι κάπω δύσκολο να παρακολουθώ όλα αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό ζητώ συγγνώμη αν δεν παρακολούθησα πολύ καλά την μέχρι τώρα συνεδρίαση. Η κυρία Χάρκιν θα με διορθώσει, φαντάζομαι, αν κάτι λησμονήσω από τα όσα έχω να πω. Ε, Καταρχά, λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό από πλευρά Σάλτε να ε, φροντίσουμε να μην κάνουμε μόνο παράπονα για την κατάσταση των γυναικών, αλλά να προτείνουμε συγκεκριμένες λύσεις για τη διέξοδο από τη φτώχεια. Ε, αυτή ήταν και η προσπάθειά μα. Για τι συμβαστικέ ε, τροπολογίε μπορούμε να δεχθούμε την υπαριθμόν Α όπω έχει. Στη Β υπάρχουν κάποιε δυσκολίε, το ακούσατε άλλωστε νομίζω. Υπάρχει μια τροπολογία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο με τον όρο τη κοινωνική ενσωμάτωση, inclusion. Και αν γίνει δεκτή αυτή η αλλαγή ορολογίας δεν έχουμε ε, αντίρρηση, εκτός από το ότι εδώ γίνεται για άλλη μία φορά λόγος περί αυξήσεως ε, της προκοδότησης του Ταμείου για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Εδώ λοιπόν η αντίρρηση μας είναι εξής, ότι είναι πολύ καλά να έχουμε χρήματα για τα ταμεία, αλλά εδώ πέρα το να ενισχύεται το Ταμείο για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση, μήπως θα ήταν, ε, ίσως δεν είναι τόσο καλή ιδέα όσο το να ενισχυθούν άλλα ταμεία τα οποία έχουν διαφορετική χρήση και στόχους. Το Ταμείο Παγκοσμιοποίηση για μα δεν θα έπρεπε να περιλαμβάνει τι αυτέ τι προτάσει. Θα έπρεπε να γίνεται λόγο μόνο για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αυτό προ την ε, συμβαστική τροπολογία υπαριθμών Β. Ε, και πιστεύω ότι συζητήθηκε και το τι θα γίνει εάν δεν περάσουν βαστικές τροπολογίε και πώς θα χειριστούμε τις επιμέρους λοιπέ δηλαδή τροπολογίες. Εάν παραδείγματι η Β δεν περάσει τότε οι 48 και 49 θα πρέπει να υποβληθούν σε ψηφοφορία σε τμήματα, με split votes δηλαδή. Και έτσι διαφωνούμε με το πρώτο τμήμα, διότι προτείνει μια σημαντική ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, ενώ το δεύτερο τμήμα μας βρίσκει σύμφωνος ε, στη διατύπωσή του. Επίσης, στην 42 ε, τροπολογία, θα ήθελα να πω ότι την υποστηρίζουμε, συζητήθηκε και αυτό το θέμα πιστεύω μέχρι τώρα, και η συμβαστική ε, για μας ε, σημαίνει ότι θα ακολουθήσουμε το ΕΛΚ, το Ευρωπαϊκό Λεκό Κόμμα, δηλαδή θα αντιδεχθούμε εφόσον διαγραφεί το δεύτερο τμήμα. Ιδάλλως, το θέμα περί πολιτικής για την αγορά εργασίας είναι η δική μου τροπολογία 52. Ε, τότε θα ήθελα να την ψηφίσουμε χωριστά εκεί όπου γίνεται λόγος για ενδείξεις που δείχνουν ότι ε, ε, evidence indicates that κτλ. Ε, αυτό μπορούμε, εφόσον φύγει αυτό το κομμάτι μπορούμε να δεχθούμε τη συμβαστική ε. Ευχαριστώ κυρία Γκέρινγκ. Girling. Ευχαριστώ πολύ. Μάλλον μειοψηφία είμαι. Ο συμβιβασμός, η συμβαστική τροπολογία Α προσθέσαμε τόσο πολλές προτάσεις, τόσο πολλές λέξεις που πραγματικά τελικά δεν έχει κανένα νόημα ω δήλωση. Ένα τμήμα με βρίσκει απολύτως σύμφωνη και συμφωνώ απολύτω ότι πρέπει να συμπεριληφθεί πρόσβαση στην αγορά εργασίας και στην εκπαίδευση και ε, βέβαια η ανάγκη για έναν αξιοπρεπή δύο. Με όλα αυτά συμφωνώ απολύτως αλλά ίσως θα έπρεπε να το θέσουμε πολύ πιο, με πιο οριστικό τρόπο για το πώς δηλαδή μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, να είμαστε κάπως πιο κατηγορηματικοί στη δήλωσή μας έτσι όπως είναι όμως τώρα η συμβαστική τροπολογία νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα να την υποστηρίξει κανείς. Αν υπήρχε κάτι πιο συγκεκριμένο για το πώς μπορούμε να επιτύχουμε τον αναφερόμενο στόχο θα συμφωνούσα απολύτως. Για τη συμβιβαστική τροπολογία B, το είπα και στην προηγούμενη συνεδρίαση και θα το ξαναπώ, οτιδήποτε μιλά για την αύξηση της ε, χρηματοδότησης, πρικοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ή του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σε αυτή τη φάση Τη στιγμή που είχαμε όλη τη συζήτηση για την, τη μη ρεαλιστική στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τον προϋπολογισμό όταν προσπαθούν τα κράτη-μέλη να τα βγάλουν πέρα, ε, δεν νομίζω ότι έχει πολύ νόημα και γι' αυτό δεν το υποστηρίζω. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. φαινόμουν να μην σα προσέχω, αλλά προσπαθούσα να δω τι μπορούμε να κάνουμε στο πλαίσιο της τροπολογία αυτή, Κοιτάξτε, από ό,τι βλέπω πρέπει να ε, τσακωθούμε πάλι με την ε, διάσκεψη των Προέδρων ε, για να δούμε τι θα γίνει με το θέμα της Επιτροπής των Γυναικών όπως είπα και στην προηγούμενη συνεδρίαση, συμφωνώ απολύτω ε, με αυτά που είπατε. Είναι απολύτως γελίο αυτό που γίνεται, αλλά είναι ένα ζήτημα που έχει ήδη εξεταστεί στη διάσκεψη των Προέδρων. Δυστυχώ, έχουμε κάποιες συμβιβαστικέ τροπολογίες, έχουν γίνει αποδεκτέ πολλέ από αυτέ από την Επιτροπή Γυναικών, οπότε πρέπει να πάμε και πάλι στην, στην διάσκεψη των Προέδρων. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν ή ό,τι μπορείτε εσείς να κάνετε για να μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτή τη διαδικασία, α ενώσουμε τις δυνάμει μα για να μπορέσουμε να, τα, να, να, να το αλλάξουμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τσίμερη και πάλι. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά και ευχαριστώ τους συναδέλφους που μίλησαν. Εδώ θα ήθελα να πω ότι είναι προφανές πως υπάρχει κάποια παρεξήγηση ως προς τα ονόματα, γιατί εγώ είχα υπόψη να θα μιλούσε η κυρία Κορνέλισεν, αλλά στην εκφώνηση του ονοματός της ακούστηκε Λόπες Φοντάνιε. Εξού και δεν μπορούσα να παρακολουθήσω ποιος μιλάει. Γιατί ήταν ξεκάθαρο ότι μιλούσαν οι πράσινοι, αλλά είχα όνομα από άλλη ομάδα, εν πάση περιπτώσει. τελικά μπόρεσα να ξαναβρω το δρόμο μου και να καταλάβω ποιος λέει τι. Είχα πει εξ αρχής ότι σε σχέση με τι ε, παρατηρήσει που άκουσα για τις συμβαστικέ τροπολογίε. ιδιαίτερα για τη ΒΕΤΑ. Θα επαναλαμβάνω και όσοι ήρθαν με κάποια καθυστέρηση και δεν να παρακολουθήσουν όλε τι συνεδρίε. Θεωρώ ότι είναι... Ε, μέχρι τώρα ε, έχει συμφωνηθεί η κοινωνική ενσωμάτωση να αντικαταστήσει τον όρο κοινωνική προστασία συμβαστική Β. Αυτό το έχουμε συμπεριλάβει στην συμβαστική μας πρόταση. Ως εκ δεν υπάρχει εδώ ανάγκη για επιπλέον τροπολογία. Άλλωστε σε αυτό έχουμε συμφωνήσει ότι δεν θα κάνουμε ε, σε τμήματα τροπολογίες στις συμβαστικές. Μπορεί κανείς να υπερψηφίσει μια συμβαστική ή να την καταψηφίσει, αλλά όχι σε τμήματα ψηφοφορία. Σε αυτό είχαμε συμφωνήσει, γιατί είχαμε πει ότι θα βρούμε μια κοινή διατύπωση και θα την υποβάλουμε σε ψηφοφορία. Αυτό λοιπόν, κοινωνική ενσωμάτωση. Τώρα έχουμε αυτόν τον όρο πλέον, ενσω... ενσωμάτωση συμπεριλάβει. Έχουμε επίσης μια, μια σαφή ε, ιδέα για το τι γίνεται με αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Η κυρία μάστη μας, είπε, μας είπε εκ μέρους της Άλντο ότι δεν θέλει να δεχθεί αυτή την ενίσχυση, την πρόταση. Τότε κοιτάξτε να σας πω. Να δηλώσω για άλλη μια φορά και κυρίως ε, για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες ότι εγώ δεν συμφωνώ ιδιαίτερος γιατί και εγώ, συμφωνώ, και εγώ βλέπω ότι είναι ε, δύσκολο να συμπεριληφθούν στο ίδιο κείμενο τα δύο ταμεία. Θα ήταν καλύτερο να τα διαγράψουμε τελείως, να μην αναφέρουμε δηλαδή ρητά τα δύο ταμεία. Είχα πει να ξανασυστήσουμε την ιδέα τη συμπερίληψη του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση, αλλά σε αυτό αντέδρασαν οι πράσινοι που δεν ήθελαν να διαγραφεί. Εν πάση περιπτώσει όμω, εγώ θα ήθελα να πείσω την κυρία Μάισνερ ε, να ακολουθήσει τη συμβαστική μα ε, τροπολογία. Γι' αυτό παρακαλώ για άλλη μια φορά, ε, μετά το τέλο τη συνεδρία, μετά το τέλο αυτή τη συζήτηση, να συζητήσουμε με του και συγκητέ και να ενημερώσουμε μετά τη γραμματεία εάν παραμένει αναφορά στο Ταμείο για την, για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση ή όχι. Για το ε ευχαριστώ πολύ όλους όσοι έλαβαν το λόγο. Ακολουθούμε νομίζω την ίδια κατεύθυνση με την επιχειρηματολογία μας. Η τελευταία φράση κλείνει με το, τους, τα, τόσο τα έσοδα όσο και τις δαπάνες. Και εκεί έχουμε τελεία και παύλα. Σε αυτό δεν υπάρχει λοιπόν ζήτημα. Το άλλο κομμάτι έχει αποσυρθεί από την συμβαστική τροπολογία και έτσι δεν πρόκειται να ψηφιστεί. Κατά τα άλλα, παρακαλώ να είμαστε σαφείς για το τι σημαίνει ενισχυμένη συνεργασία. Είναι καλό να είναι ξεκάθαρη κατάσταση και με τη διάσκεψη των Προέδρων να ε, γίνει η σχετική διαπραγμάτευση για να διευκρινιστεί το θέμα αυτό. Εξού και εγώ θα πρότεινα να μην επιδιώξουμε πλέον στην υπόθεση αυτή την ενισχυμένη συνεργασία όπως τη λέμε διότι θα πρέπει να προσδιορίσουμε εμείς, να χαράξουμε εμείς το δρόμο για να ξέρουμε προς τα πού πηγαίνουμε. Και από εκεί και πέρα καταθέτουμε τροπολογίες, τις υποβάλλουμε στην Επιτροπή των Γυναικών και εφόσον θέλει τις δέχεται. Έχουμε αυτή την ιστορία με τις ε, αρμοδιότητες των δύο επιτροπών, ε, την οποία βρίσκουμε μπροστά μας δυστυχώς κάθε φορά. Ε, δεν είναι εύκολο να κάνουμε μια έκθεση μόνο εάν δεν την έχει αναλάβει η Επίτροπη των Γυναικών. Η Επιτροπή των Γυναικών και πέρας περιπτώσει δεν είμαστε και παράρτημα της Επιτροπής των Γυναικών. Δεν μπορούμε να το δεχθούμε αυτό. Αυτό. Κατά τα άλλα, να έχουμε καλύψει πιστεύω τα κύρια ζητήματα. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά ως συναδέλφους έλαβαν τον λόγο. Ευχαριστούμε, κυρία Ζήμερη. Η ψηφοφορία, που ξέρετε, είναι αύριο το πρωί στις 9.30. Και περνάμε στην επόμενη έκθεση. Να δώσω το λόγο απευθείας στην κυρία Χάρκιν. ΑΕΠ και επέκεινα. Καταμέτρηση της πρόοδου σε έναν μεταλλασσόμενο κόσμο. Κυρία Χάρκιν, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους όσοι υπέβαλαν τροπολογίες Με μεγάλη μου χαρά πρέπει να πω ότι πολλές τροπολογίες έχουν βελτιώσει αισθητά το κείμενο. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στους συναδέλφους. Προσπάθησα να συμπεριλάβω όσο το δυνατόν περισσότερες συμβαστικέ τροπολογίες. Υπάρχουν κάποιες άλλες που τις σημείωσαμε πλην στην, ε, στο κατάλογο των ψηφοφοριών, όχι γιατί διαφωνώ με τις τροπολογίες αυτές καθεαυτές, αλλά γιατί νομίζω ότι η έννοια, η ιδέα που εξέφραζαν ήδη περιλαμβανόταν στις συμβαστικές τροπολογίες στο υπάρχον κείμενο. Προσπάθησα να βεβαιωθώ ότι η έκθεση θα είναι συνεπής και ότι λόγω χάρη δεν θα επαναλάβουμε το ίδιο πράγμα δύο φορές. Ως γενική παρατήρηση πρέπει να πω για το θέμα του ΑΕΠ και επέκεινα ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε συνεπή δράση. Και ενώ υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία καλύπτει η δική μου γνωμοδότηση, πρέπει επιπλέον να γνωρίσουμε ότι σε κάποια σημεία θα πρέπει να έχουμε μια κοινή αντιμετώπιση και να δούμε τι αντίκτυπος θα υπάρχει στην πολιτική μας. Τι είναι μια γενική παρατήρηση. Από την άλλη αναγνωρίζουμε την ανάγκη να πάμε πέρα από το ΑΕΠ και ότι υπάρχουν επιπλέον δείκτες που πρέπει να συμπεριληφθούν. Είμαι λοιπόν ιδιαίτερα ικανοποιημένη με την τοποθέτηση που εκφράζεται εδώ. Όπω είπα, υπάρχουν διάφορε τροπολογίε και κατάλογοι και προσπάθησα κάποια ζητήματα να τα καλύψω μόνο μία φορά. Άλλαξα τον όρο measure, ε, μέτρηση, σε δύο σημεία για να μπει στη θέση του οι δείκτες. Αυτό ήταν σημαντικό για κάποιους συναδέλφους και το έκανα με ιδιαίτερη χαρά. Επίσης, ένα σχόλιο για την τροπολογία 57. Υπάρχει ένα σφάλμα εκεί. Για την τροπολογία 57 δεν περιλαμβάνεται. Το συζητήσαμε με την κυρία Τίμερ, το γνωρίζει ακόμη όμως παραμένει στον κατάλογο των ψηφοφοριών. Δεν θα συμπεριλαμβάνεται στην συμβαστική ΑΕ και θα ψηφιστεί ξεχωριστά. Συγγνώμη, κυρία Χάρκιν, να σα διακόψω και να πω ότι όσοι συζητούν ακόμη σε πηγαδάκια για την προηγούμενη έκθεση, αν μπορούν να το κάνουν αυτό εκτό αιθούση. Είναι πολύ ενοχλητικό για όσου προσπαθούν να εργαστούν επ' αυτή τη έκθεση. Κυρία Ζήμερ, μπορείτε να συζητήσετε εκτό αίθουσα. Ενοχλείτε όσους προσπαθούν να ακούσουν αυτή τη συζήτηση. Κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ. Σχεδόν ολοκλήρωσα. Υπάρχει ένα ζήτημα που θέλω να θίξω εδώ. Το συζήτησα και με τον κύριο Ντόιτ, είναι η τροπολογία 64, η οποία αναφέρει το ΑΕΠ ως βασικό κριτήριο για να ορίσουμε την επιλεξιμότητα για τις περιφερειακές ε, πολιτικές και Εδώ ένα μέρο τη τροπολογία μιλάει για εθνικέ αρχέ που δίνονται να εφαρμόζουν στο κατάλληλο επίπεδο λήψη αποφάσεων άλλου δείκτε. Εδώ ξέρω ότι υπάρχει θέμα στην Επιτροπή Ρέτζι των Περιφερειών και θα πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία και εκεί, οπότε και εμεί θα πρέπει να, συντονιστούμε για να δούμε αν θα μιλήσουμε για σημαντικό κριτήριο ή για βασικό core κριτήριο. Διότι αν πιστεύουμε ειλικρινώς όπως λέει η πρώτη συμβαστική τροπολογία, ότι το ΑΕΠ είναι σημαντικός μεν δείκτης για την οικονομική ανάπτυξη, αλλά είναι πλέον ε, κατάλληλο ως μοναδικό εργαλείο για να καθοδηγεί το σχεδιασμό πολιτικών. Ε, νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση είναι λογικό στην συνέχεια της έκθεσης να λέμε ότι για αυτό το συγκεκριμένο τομέα το ΑΕΠ θα μπορούσε να παραμένει το μόνο κριτήριο. Και για τις ε, περιοχέ του στόχου 2 υπάρχουν και άλλοι δείκτε που ήδη χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν την επιλεξιμότητα. Νομίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε για το σημείο αυτό, να κάνουμε πιο ήπια την έκφραση και να παραμείνουμε στην βασική ιδέα τη έκθεση πιστή. Ε, θέλω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσω τι απόψει των συναδέλφων. Να, σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριος Χώμα. Good heavens, thank you, Madam Chairman. astonished to be first. Ευχαριστώ. Πραγματικά μου κάνει πολύ εντύπωση που παίρνω πρώτος το λόγο για το ΕΛΚ σήμερα. Έχουμε σοβαρές ανησυχίες. Σηκώσατε πρώτο το χέρι, γι' αυτό σας έδωσα το λόγο πρώτο, γι' αυτό πήρα το λόγο πρώτος, λέει η Πρόεδρος. Μάλιστα, μεγάλη σας καλοσύνη. Λοιπόν, έχουμε σοβαρές ανησυχίες ε, για την έκθεση αυτή. Το θέμα είναι ότι το ΑΕΠ ε, είναι ένας ε, παγιωμένος ε, και πολύ είναι ένα πολύ παγιωμένο μέτρο, αντικειμενικό, πολύ γνωστό, χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο, ε, είναι εύχριστο για διεθνείς ε, συγκρίσεις και ακούω διάφορους εδώ στην αίθουσα που λένε ότι αν ναι, ε, είναι αρκετά σημαντικό σε αυτός ο δείκτης, όμως έχω την εντύπωση ότι ο στόχος της έκθεσης είναι να περιθωριοποιήσουμε το ΑΕΠ και να συμπεριβάλλουμε άλλους δείκτες. Και νομίζω ότι παραγνωρίζοντας έναν πολύ εύχριστο, πολύ κατανοητό και πολύ α, αντικειμενικό μέτρο Υπάρχει μια τάση, ειδικότερα στη δική μας Επιτροπή, να, εισα, να εισαγάγουμε άλλους δείκτες, λιγότερο αντικειμενικούς, ε, βάσει διάφορων ε, ε, ιδεολογικών απόψεων και όχι βάσει τοποθετήσεων που βασίζονται σε συγκεκριμένα στοιχεία πιο αντικειμενικά. Όσον αφορά τους νέους οικονομικούς δείκτες στην τροπολογία 31, κοιτάξτε, εμένα αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ ε, μυστήριο αίτημα. Πρέπει να μας πείτε ποιοι είναι αυτοί οι δείκτες. Επίσης ζητάτε αντικατάσταση του ΑΕΠ ε, ως βασικότερου δείκτη ε, καθορισμού της πολιτικής. Ε, επαναλαμβάνω λοιπόν αυτά που είπα, ότι αυτός ο δείκτης είναι ευρέως αποδεκτός σε όλο τον κόσμο και δεν ξέρω αν κανείς έχει καμιά καλύτερη ιδέα για ένα νέο τέτοιο δείκτη. Εντάξει, υπάρχουν πολλοί οικονομικοί δείκτες. Ε, η ανησυχία που έχω είναι μήπως θα έπρεπε να πάρουμε αυτόν το δείκτη ο οποίος είναι ο πιο γνωστός και πιο αντικειμενικός. Και τούτου λεχθέντος έχω να προτείνω το εξή έχουμε μία κατάσταση εντός της Ευρωζώνης, που τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης ε, έχουν απολέσει την ικανότητά τους ε, να επηρεάσουν την νομισματική τους πολιτική και τα επιτόκια τους και βλέπουμε κάποιες χώρες όπως η Ελλάδα, αλλά όχι μόνο η Ελλάδα, που πάρα πολύ υποφέρουν από την κατάσταση αυτή. Αν θέλουμε λοιπόν επιπλέον οικονομικούς δείκτες, ίσως θα έπρεπε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφεύρει έναν οικονομικό δείκτη που θα μετρά την ε, ζημιά που κάνει το ευρώ στην, ε, στις χώρες ευρωζώνης. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Λάμπερτ και μετά η κυρία Μωρέν Σαρτιέ. Πρόεδρε, <clears throat> θέλω να ευχαριστήσω την εισηγητρία που καλωσόρισε τα σχόλιά μας και τον κύριο Χάλμερ που μίλησε για τις τροπολογίες 41 και 45, διότι εδώ θίγονται ζητήματα χρονοδιαγράμματος για το πώ θα περάσουμε από το ένα σύνολο δικτών στο άλλο. Είναι σημαντικό λοιπόν και είναι σαφή εδώ η έκθεση. Το έργο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο παρελθόν, το έργο του Ευρωκοινοβουλίου από το παρελθόν και τη βρετανική κυβέρνηση μάλιστα από το παρελθόν, ε, των συντηρητικών δηλαδή, ε, εκεί που έγινε μια αναζήτηση νέων δικτών, είναι πολύ σημαντικό. Η ανησυχία πολλών από εμά με το ΑΕΠ είναι ότι όπως ε, και η κυρία Χάρκιν πολύ σαφώς τον τοπίζει στην έκθεση, από το να είναι απλό οικονομικό δείκτης τίνει να γίνει ο, πλέον, ο κατεξοχήν στόχος. Ε, είτε πρόκειται για τα στατική της Λισαβόνας και για άλλου τομεί. Ιδίω για μέτρα αύξησης ε, του ΑΕΠ, τα οποία πάντοτε κρίνονταν ω Δεν συνεξετάζαμε όμως και τον αντίκτυπο που θα είχε ε, η παροχή περισσότερων χρημάτων ε, στην ε, οικονομία, τι γίνεται με τη δαπάνη των ε, κονδύλιων. Και ένα κλασικό παράδειγμα είναι ότι μπορεί να είναι πολύ καλές για το ΑΕΠ οι πετρελαϊκές δραστηριότητες και η χρήση, ο καθαρισμός μάλλον, αλλά δεν είναι απαραίτητος καλή η χρήση του πετρελαίου για το περιβάλλον, για την ποιότητα ζωής. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποιοι άλλοι δείκτες μπορεί να υπάρχουν που να δώσουν δυνατότητα για διαφορετική μέτρηση και μια πιο πλήρη συνολική εικόνα. Να μην ε, επαφιόμαστε πλήρως όπως έκαναν τώρα πολλές ε, πολιτικές και οι πολιτικοί θύνοντες βεβαίως στο ΑΕΠ που θα είναι το κατεξοχήν ε, μέτρο σύγκρισης για την πρόοδο. Είναι περιορισμένη, είναι κοντόφθαλμη αυτή η προσέγγιση. Όσο για την τροπολογία 45, αυτό που ζητούσαμε εδώ είναι να αντικατασταθεί ο το ΑΕΠ ως πλέον σημαντικός δείκτης, ως βάση λήψη αποφάσεων για όλου των ειδών των αποφάσεων που δεν σχετίζονται παρατήτως με την περαιτέρω παροχή κονδυλίων σε ένα συγκεκριμένο τομέα της οικονομίας. Νομίζω λοιπόν ότι η κατεύθυνση τη έκθεση τη κυρία Χάρκιν είναι πολύ θετική. Θα στηρίξουμε τι τροπολογίε και συμφωνούμε με τι ανησυχίε τη για την τροπολογία 64. Ελπίζουμε ότι θα βρούμε εδώ μια εναλλακτική διατύπωση και θα ήμασταν ιδιαίτερα ευγνώμονε αν το πετυχαίναμε αυτό. Ιδάλω θα την καταψηφίσουμε. Ω προ τι υπόλοιπε τροπολογίε που έχουν υποβληθεί, ε, ίσως να μην ταιριάζουν όλες με, τη, με μια έκθεση περιδικτών δεν επικεντρώνονται στο ίδιο θέμα όπως η έκθεση. Αυτό είπε και η κυρία Χάκινγκ. Ελπίζω λοιπόν ότι θα καταλάβετε από την στάση μα την αυριανή ψηφοφορία ότι αν καταψηφίσουμε κάποιε τροπολογίε είναι επειδή θέλουμε να παραμένουμε πιστοί στην κεντρική ιδέα τη έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μωράν Σαρτιέ. Και μετά κυρία Μωράλε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ήθελα καταρχά να αποκτήσω φορό τιμή στο έργο τη κυρία Χάρκιν η οποία εργάστηκε όπως το συνηθίζει με πολύ ευσυνειδησία. Βλέπουμε ότι από τότε που άρχισε να χρησιμοποιείται η έννοια του ΑΕΠ, τα πράγματα έχουν αλλάξει, θα πρέπει να προχωρήσουμε κι εμείς και στην αντίληψή μας του ίδιου του ΑΕΠ. Ωστόσο, πρέπει να σας πω εξ ονόματος του ΕΛΚ και το λέω και στον κύριο Χέλμερ που ανησυχούσε για τη στάση του ΕΛΚ, πρέπει να πω ότι κάποιοι από τους συναδέλφους μου ανησύχησαν ότι κάποια από τα κριτήρια που προτείνονται μέσω των τροπολογιών που σήμερα βλέπουμε να έχουν υποβληθεί, κάποια από αυτά τα κριτήρια δεν είναι αρκετά μετρήσιμα δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μελετών ε, για τον αντίκτυπο που θα έχουν όλα αυτά που προβλέπουμε σε σχέση με τις πολιτικές αποφάσεις που θα προξενήσουν, στις οποίες θα βασιστούν. Κάποιοι δείκτες αφορούν άμεσα τη ζωή των, την ίδια των πολιτών. Ε, και μάλιστα την πολύ, το πολύ προσωπικό βίο των ε, πολιτών. Τον ιδιωτικό τους βίο σχετίζονται με συστήματα που είναι πολύ δύσκολο να μετρηθούν, να καταμετρηθούν με τρόπο αντικειμενικό. Αυτό είναι και ο λόγος που λόγω χάρη οι δείκτε για τον ειδικό βίο, για, για την νοητική ευζοία, βλέπουμε ότι μπορεί σε ένα κράτος να υπάρχει ένα πολύ ψηλό ΑΕΠ, αλλά άνθρωποι που έχουν πολύ χαμηλό επίπεδο ζωής, διότι η χρήση η χρήση των όσων αποφέρει το ΑΕΠ δεν τίθενται στην υπηρεσία τους. Από την άλλη, βλέπουμε ότι κάποιες προτάσεις για νέους δείκτες είναι ιδιαίτερα αμφισβητήσιμοι. Ε, στέκονται σε σημεία πολύ ευαίσθητα και θα είναι εξίσου ευάλωτη και η στατηγική ανάλυση τους. Γι' αυτό αρκετοί από τους συναδέλφους μου ανησύχησαν με αυτές τις προτάσεις, γι' αυτό σήμερα δεν θα συμφωνήσω με τη συμβαστική τροπολογία C, D, Ε και F που προτείνουν ακριβώς αυτούς τους δείκτες που είναι ιδιαίτερα αμφισβητήσιμοι, ευάλωτοι και δεν μπορούμε να τους καταμετρήσουμε, δεν είναι σταθεροί. Αυτή είναι η θέση του Ελκενολίγης. Ακόμη και αν γνωρίζουμε καλά ότι πρέπει να εξελιχθεί η έννοια του ΑΕΠ. Πρέπει να εξελιχθεί. Και να βασιστεί σε δείκτες σταθερούς, μετρήσιμους, που να μπορεί κανείς να τους αντιληφθεί εύκολα και να τους χρησιμοποιήσει. Αλλά να γίνει και μια χρηστή αξιοποίησή τους. Ευχαριστούμε. Κύριε Μοράλης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ χρήσιμη και πολύ έγκαιρη αυτή η έκθεση και λόγω της ε, κρίσης ε, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε πολύ ακριβείς και πολύ ε, ενημερωμένες στατιστικές έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν σοβαρές κοινωνικές συνέπειες, αλλά δεν ε, υπήρξε κανένας δείκτης που να λέει κάτι περισσότερο για την κοινωνική αυτή κρίση. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, χρόνο για να το επεξεργαστούμε και θα ήθελα να ζητήσω από όσους λένε ότι το ΑΕΠ είναι πολύ σημαντικός δείκτης. Είναι γεγονός, αλλά και κάτι που καλύπτει πολλές από τις ε, διαδικασίες που έχουν να κάνουν ε, με την ανισότητα, με ε, την αύξηση της φτώχειας, με τις διαφορές που υπάρχουν στις διάφορες χώρες μέλη. Αυτό όμως που αναφέρουμε στις ε, τροπολογίες είναι ότι πρέπει να εργαστούμε επί, την, επί των πτυχών αυτών ε, της ε, ανάπτυξης των συνθήκων εργασίας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ληφθεί υπόψη λοιπόν όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί το, λόγω των αλλαγών. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ την κυρία Χάρκιν για την δουλειά της. Είναι πάρα πολύ καλές οι συμβιβαστικές τροπολογίες και πραγματικά έχουν καταφέρει να συγκεράσουν ε, τις ε, ε, διαφορετικές προτάσεις και μπορούμε έτσι να καταλήξουμε σε κάτι σημαντικό για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τσίμερ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Χάρκιν για τη δουλειά της είχαμε πει ότι θα γίνει μια συζήτηση για αυτό το θέμα του ΑΕΠ και την ε, μέτρηση της πρόοδου. Να δούμε δηλαδή τι μπορεί να σημαίνει από απόψε ως ε, ανάπτυξης και ε, οικολογίας, για παράδειγμα. Οι περισσότερες τροπολογίες που υπέβαλε η, ομάδες, η ομάδα μου έχουν συμπεριληφθεί στις συμβιβαστικές τροπολογίες, αλλά δυστυχώς το αίτημά μας για τη μέτρηση της προόδου για να η τροπολογία μας που αφορά ειδικότερα τη μέτρηση της προόδου δυστυχώς δεν συμπεριλήφθηκε. Πρέπει να πω όμως ότι βάσει των τροπολογιών αυτών είναι πολύ πιο πλήρης η έκθεση και επομένως μπορούμε να υποστηρίξουμε τις συμβιβαστικές τροπολογίες εκτός από την υπαριθμόν 1 γιατί εκεί δεν έχουμε συνδυάσει, δεν, δεν έχουμε συνδυάσει το θέμα με την καλή ποιότητα εργασίας. Ευχαριστούμε λοιπόν για τη δουλειά σας, κυρία Χάρκιν. Η κυρία Σρέτε, Εγώ θα ήθελα να επανέλθω στην πρώτη παρέμβαση που αφορούσε το γεγονός ότι το ΑΕΠ ε, δεν μας ε, οδηγεί στο σωστό αποτέλεσμα στις πρώτες προτάσεις είναι απολύτως σαφές ε, ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά και ότι δύο τρίτα των πολιτών ε, νιώθουν ε, την κακή κατάσταση που υπάρχει. να μην ξεχνούμε και ε, όλα αυτά που υπόθηκαν σε επίπεδο όσα Είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά και την κυρία Χάρκιν, αλλά και την ε, προσπάθεια ορισμένων ε, που προέρχονται από τον αριστερό πολιτικό χώρο να εφεύρουν κάτι είναι γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με κάτι το οποίο είναι σαφέστατα αναγνωρισμένο, όπως είναι ο δείκτης του ΑΕΠ, Όμως για μένα το σημαντικότερο τμήμα της ανακοίνωσης είναι ότι δεν υπάρχουν ε, εμπόδια που δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε όταν θέλουμε να περιγράψουμε μία κατάσταση που αφορά το κατά πόσο σημειώνει πρόοδο μία περιφέρεια ή όχι. Επομένως, το Κοινοβούλιο στη συντριπτική του πλειοψηφία, στην περασμένη Ολομέλεια, ψήφισε το ότι πρέπει να συμπεριληφθούν και άλλου είδους δείκτες πέρα από το δείκτη του ΑΕΠ γιατί είναι κάτι το οποίο δουλεύει και σε εθνικό επίπεδο. Μπορούμε να συμπεριλάβουμε και άλλους δείκτες πέρα από το ΑΕΠ και, που μπορούμε, και μπορούμε έτσι να περιγράψουμε καλύτερα την ε, κατάσταση σε μία περιφέρεια και το γεγονός ότι υπάρχουν ε, διαφορές ε, στο ε, εισόδημα κάποιων ανθρώπων δεν είναι απαραίτητος και δείκτης του τι πρέπει να γίνει προκειμένου να σημειωθεί πρόοδο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός λοιπόν ότι πρέπει να εξετάσουμε το ζήτημα αυτό πιο προσεκτικά και να καταλάβουμε κάτι το οποίο είναι απολύτως σαφές πλέον στους περισσότερους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι γεγονός ότι το ΑΕΠ δεν επαρκεί ως δείκτης μέτρησης. Ο κύριος Ευχαριστώ. το ΑΕΠ δεν είναι ο τέλειος δείκτης, σίγουρα. Όμως πρέπει να προσθέσω ότι είναι και ένα αντικατάστατο. Γιατί, διότι ακριβώς καταμετρά κάτι. Τι ακριβώς μετρά, την οικονομική δραστηριότητα ετησίως. Εάν με επιτρέπετε, θα προσπαθήσω να ανακαλύψω μαζί σας τι γίνεται με τα 14-15 κριτήρια που έχουμε μπροστά μας και τι καταμετρούν. Να αναφέρω ορισμένα. Η εγκληματικότητα, η πολιτιστική συμμετοχή, η οικογένεια το επίπεδο της εμπιστοσύνης του κοινού. Το mental well-being, η ευζοία, η νοητική, ας το αφήσω στα αγγλικά. Ε, γιατί να μην προσθέσουμε και την κοινωνική διαδικτύωση, στο social networking σε αυτή τη συλλογή. Κοιτάξτε, είναι πολύ συγκεκριμένε οι τροπολογίες και δεν θα ήθελα να περάσετε στις λεπτομέρειες. Αν θέλετε να πάτε στα σημαντικά σημεία, ε, τα βασικά σημεία των τροπολογιών, δεν γίνεται τώρα να διατρέξουμε 40 τροπολογίες. Πολύ καλά, κατάλαβα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σχολιάσω λοιπόν την τροπολογία 4, η οποία ε, διατυπώνει, διαγγέλει μάλλον, ευθύ εξ αρχή ότι είναι παροχημένο και ακατάλληλο ο δείκτη του ΑΕΠ. Νομίζω ότι σε μια σοβαρή οικονομική συζήτηση μια τέτοια δήλωση δεν έχει θέση. Επίσης η τροπολογία 17, ε, αντικειμενική ε, ευζοία, υποκειμενική μάλλον ε, ζωή. Αυτό είναι κάτι που έχει σχέση και με την τροπολογία, τη συμβαστική τροπολογία C και είναι και τελείως υποκειμενικό. Ευχαριστούμε. Η κυρία Χάρκεν για να ανακεφαλαιώσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα ίσω να σχολιάσω κάποια από τα ζητήματα που εφήγησαν. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Χέλμερ. Είναι ένα καταξιωμένο δείκτη το ΑΕΠ, Όμω, πιστεύω ότι οι περισσότεροι εδώ συμφωνούν. Χρειαζόμαστε επιπλέον δείκτε και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει πει. Και παραθέτω, είναι μια σαφή περίπτωση, διαφαίνεται η ανάγκη συμπλήρωση του ΑΕΠ με άλλου οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού δείκτε. από του οποίου εξετάται άμεσα η ευζοία των ανθρώπων. Εδώ λοιπόν το θέμα δεν είναι να χρειαζόμαστε επιπλέον δείκτε, αλλά το ποιου θα διαλέξουμε. Και το είπα αυτή εξ αρχή, ότι χρειάζεται να είμαστε συνεπεί ω προ του εαυτού μα. Ε, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι το ΑΕΠ λόγω χάρη δεν μετρά την περιβαλλοντική ιδιωσιμότητα. Αν θέλουμε τώρα να αποψηλώσουμε όλα τα δάση στην Νότια Αμερική, αυτό θα αυξήσει το ΑΕΠ. Όμω δεν θα κάνει και πολλά για το καλό του περιβάλλοντο. Σωστά. Ε, ε, ο αριθμό των ε, φυλακών επίση έχει αυξηθεί εντυπωσιακά. Εάν γίνει κάτι τέτοιο και συνεχιστεί αυτή η τάση, θα αυξηθεί το ΕΠ, αλλά δεν θα βοηθήσει τίποτα αυτό την κοινωνία του πολίτε. Νομίζω λοιπόν ότι όλοι συμφωνούν ότι υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω δείκτε. Νομίζω ότι αρκετά τα είπαν ήδη οι δεν θέλω να τα επαναλάβω και δεν θα επιμείνω σε αυτό. Απλώς να πω στην κυρία Μωράν Σαρτιέ ότι είχα την αίσθηση ότι σε κάποιες από τις εμβαστικές τροπολογίες που αναφέρατε είχα ήδη καλύψει τις ανησυχίες σας προσθέτοντας τους όρους λόγου χάρη. Δείτε τις F και G. Μιλώ για τις διαφορετικές κατηγορίες, αλλά δεν έδωσα έναν απλό κατάλογο. Χρησιμοποίησα το επιπαραδείγματι, το λόγο χάρη, για να φανεί ότι υπάρχει επιλογή εδώ. Υπάρχουν πολλέ επιλογέ μεταξύ των οποίων μπορούμε να διαλέξουμε. Όπω, η φτώχεια και η πολιτιστική συμμετοχή πολλέ από αυτέ ε, προτάθηκαν από μέλη του ΕΛΚ. Αντί λοιπόν να αποφασίσουμε ποιε θα είναι οι διάφορε κατηγορίες συγκεκριμένα, εγώ προσπάθησα να συμπεριλάβω στου δείκτες μου φαίνονταν λογικοί, συμπεριλαμβάνοντας το λόγου χάρη, ενδεικτικά. Δηλαδή ότι η επιλογή θα πρέπει να γίνει αργότερα. Νομίζω ότι είναι λογικό αυτό και ότι μάλλον θα μπορούσαμε να βρούμε κάποιο είδου συνεννόηση και συμφωνία. Αλλά έχουμε ήδη προχωρήσει αισθητά προ αυτή την κατεύθυνση. Κυρία Τσίμερ, ναι. Καταλαβαίνω τι λέτε. Αυτό μπορούσαμε να κάνουμε τις συμβαστικές τροπολογίες και όχι κάτι παραπάνω. Επίσης ο συνάδελφος που μίλησε για την ανάγκη να προσθεθούν δείκτες και ο κύριος Άγγλ που είχε δίκιο για την τροπολογία 4. Αν δείτε βέβαια την τροπολογία 5 που είναι δική μου, την έχω αλλάξει. Μάλλον έχω αλλάξει εγώ ίδια το κείμενο, το total, το πλήρως. Το έχω φροντίσει να διορθωθεί. Και για το 17 δεν πρόλαβα να το δω ακόμη, αλλά εδώ έχουμε την τροπολογία της κυρίας Γκάνης. Συμφωνώ η κάθετη διανομή δεν είναι απαραίτητα ε, το ευκταίο και αν δείτε συνολικά το θέμα της διανομής σίγουρα είναι σημαντικό αλλά δεν είναι απαραίτητο να ε, γίνεται σε κάθετη βάση. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ψηφίσουμε αύριο για το θέμα αυτό και πάλι στις 9.30. Τώρα έχουμε να δούμε την υλοποίηση των οδηγιών για τις υπηρεσίες και η συγγήτρια είναι ο κύριος, η συγγητής μάλλον ο κύριος Μπεναμίας, Ζαναλίου Μπεναμίας. Και ας μιλήσουν δύο λεπτά όλοι εκτός από τον εισηγητή. Προσπάθησα να είμαι όσο το δυνατόν πιο συνοπτικός. για μια οδηγία αρκετά ευαίσθητη και που επιζητά συμβιβασμούς ε, όπως αυτούς που θα σας προτάνω. Για την παράγραφο 1 υπάρχει συμβιβαστική τροπολογία όσον αφορά το συμβιβασμό C, γ. Ξαναέγραψα τις τροπολογίες 16, 17 και 18. Μάλλον δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα αυτό σε καμία πολιτική ομάδα. Όσον αφορά την παράγραφο 2, συμβιβαστική δέλτα. D. Τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα. Προτείνω ένα συμβιβασμό των τροπολογιών 23, 24, 28 και 29. Παράγραφος 4 που δημιουργεί τα περισσότερα προβλήματα. Δεν υπάρχει συμβιβασμός επ' αυτού. Πρέπει να πω ότι η προφορική τροπολογία του κυρίου Μπαλτασάρ μου φάνηκε κατά κάποιο τρόπο συμβιβαστική και νομίζω ότι ανταποκρίνεται στις δηλώσεις του Επιτρόπου Μπαρνιέ για το θέμα αυτό. Για την παράγραφο 5, συμβιβαστική Ή. Προσπάθησα να συμβιβάσω τις τροπολογίες 41 έως 44. Και για την παράγραφο 6, συμβιβαστική F, σίγμα ταφ τροπολογίες 50, 51, 52, 53, 54 και 55. Περνάμε τώρα στις αιτιολογικές σκέψεις. Συμβιβαστική Α για τις τροπολογίες 2, 4 και 5. Συμβιβαστική Β για το Α, τροπολογίες 8 και 9. Νομίζω ότι αναφέρθηκα σε όλους τους συμβιβασμούς. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν δυσκολίες, τις κατανοώ και ειδικότερα στην παράγραφο 4, το ξαναλέω. Ευχαριστώ πολύ, Ελίζα Μπεθσρότερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η σκιώδη συγκήτρια που διαπραγματεύτηκε με το. Ω σκιώδη μάλλον που διαπραγματεύτηκε με τον Ζανλίκ θα ήθελα να παρουσιάσω και εγώ κάποια σχόλια. Εκ μέρου τη συναδέλφου. Υπάρχουν πολλέ τροπολογίε με τι οποίε συμφωνούμε και μπορούμε να τι στηρίξουμε. Γενικά για την νομική βεβαιότητα συμφωνώ με την κατεύθυνση που ακολουθεί η έκθεση, αλλά δεν ξέρουμε εάν οι ορισμοί είναι ακριβώς αυτοί που θέλουμε να... αυτοί που ανταποκρίνονται στην ε, ε, οδηγία. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, ιδίω σε μια στιγμή όπου αποφασίστηκε η... σε σχέση με την οδηγία, τη στιγμή που εγκρίθηκε η οδηγία για τις υπηρεσίες. Υπάρχουν αλλαγές υπάρχουν περισσότερα δικαιώματα πλέον για τα κράτη-μέλη. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Δεν πιστεύω ειλικρινώ ότι ένα τέτοιο ορισμός είναι πραγματικά εύχριστος. Δεύτερη παρατήρηση. καθοριστική σημασία κατά την άποψή μου. Κάτι με το οποίο συμφωνούμε πολύ με τον Ζαν για τις καλύτερες συνθήκες εργασίας. Πλήρης στήριξη σε αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί θα συμπεριληφθεί και στι συμβαστικέ. Ε, ήθελα λοιπόν επάνω στου συναδέλφου να κάνω αυτέ τι δύο παρατηρήσει και να εκφράσω τι ευχέ μου για καλή τυχαία στην ψηφοφορία. Ευχαριστούμε ο κύριος Κρίστερνσεν και μετά η κυρία Μωράν Σαρτιέ. Κύριε Κρίστερνσεν, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. κυρία Σέτερ το είπε ότι όπως και εκείνη και εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε την, τον εισηγητή για το έργο του. Νομίζω ότι οι συμβιβαστικέ τροπολογίες συμπεριλαμβάνουν όλα τα ζητήματα που πρέπει να περιλαμβάνονται παρά τους περιορισμούς που επιβάλλει η οδηγία για τις υπηρεσίες. Είναι πολύ σημαντικό από την άποψη της ελευθερίας μετακίνησης των εργαζομένων και της παροχής πληροφοριών, ε, υπηρεσιών συγγνώμη, πέρα από τα σύνορα των εθνικών κρατών, να μην υπερισχύουν ε, των δικαιωμάτων των εργαζομένων οι κανόνες της εσωτερικής αγοράς. Και αυτό έχει δημιουργήσει ήδη κάποια προβλήματα σε ορισμένα κράτη-μέλη. Αληθεύει ότι, όπω λέει και ο συγκεκριτή, υπάρχουν δυσκολίε. Στην παράγραφο 4 πρέπει να έχουμε έναν επιπλέον ορισμό. τι οι υπηρεσίε γενικού ενδιαφέροντο σημαίνουν και τι ακριβώ οι υπηρεσίε γενικού οικονομικού ενδιαφέροντο. Δύσκολο να γίνει διάκριση, δύσκολο να δοθεί ο σωστό ορισμό. Διότι τα κράτη-μέλη εισήγαγαν αυτό που θα πίστευαν ότι θα έπρεπε να εισηχθεί σε αυτού του τομεί. Όμω παραμένει ανάγκη για περισσότερη στόχευση και αποσαφήνεις του τι σημαίνουν τα ζητήματα αυτά. Ευχαριστούμε και πάλι τον εισηγητή για το έργο του. Σας ευχαριστώ κυρία Μωράν Σαρχέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με όλους όσους ε, επένεσαν ε, τη δουλειά του Ζων Λουκ για το ΕΛΚ, και θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, εμείς συμφωνούμε με τη συμβιβαστική α και β και δέχεται επίσης και τις συμβιβαστικές Σ και Ι. Εξακολουθεί να υφίσταται βέβαια το πρόβλημα με την παράγραφο 2D, η οποία ε, όπως είναι αυτή τη στιγμή δεν είναι αποδεκτή από το ΕΛΚ. Δεν συμφωνεί λοιπόν το ΕΛΚ ε, με την παράγραφο αυτή και την συμβιβαστική τροπολογία της παραγράφου αυτού και για την παράγραφο 6, για τη συμβιβαστική, 6, για τη συμβιβαστική F, συγγνώμη, ούτε με αυτή συμφωνούμε. Για την παράγραφο 25 τώρα, το ΕΛΚ έχει σοβαρές, σοβαρότατες επιφυλάξεις και ε, θεωρεί ότι η ψηφοφορία επί του ζητήματος αυτού είναι εξαιρετικά σημαντική. Αυτά λοιπόν εκ μέρου της πολιτικής μας ομάδας και τον τρόπο που θα ψηφίσουμε αύριο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γκρούνη και μετά ο κυρίος ε, Παλταζάρ. Πασκάλ Γκρούνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστώ τον κύριο Μπεναμιά. Ήταν περίπλοκο το θέμα το οποίο έλαβε να επεξεργαστεί. Και θα ήθελα μόνο να κάνω μια ερώτηση για την τροπολογία 46 που έχω καταθέσει εγώ, που λέτε ότι προτιμάτε να καταψηφιστεί. Ενώ στόχο έχει να βοηθήσει τους, τους πολίτες ώστε να έχουν μια καλύτερη ορατότητα, δηλαδή να μπορούν να βλέπουν καλύτερα το τι συμβαίνει. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Uh, Mr. Ευχαριστώ κύριε Βαλτασάρη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν έχω και πολλά να προσθέσω πέραν των όσων είπε η συνάδελφος εκ μέρους του ΕΛΚ. Απλώς αισθάνομαι ότι είχα το, το καθήκον όφυλα να... να εκφράσω την ικανοποίησή μας για το έργο του συγκεκριμένου. πραγματικά πάσχησε για να βρει σε μια Συμφωνία και συνεννόησης για να είμαστε συνεπείς στην προσέγγιση ενό θέματο ιδιαίτερα επίκαιρου. Πάντως το κομβικό σημείο είναι παράγραφος 4. Εκεί είναι δύσκολο να φανταστούμε ότι θα μπορέσουμε να συγκλίνουμε τελικά. Διότι υπάρχουν ε, και άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί από άλλου συναδέλφου. που αλλά αλλάζουν κάπως το πνεύμα της προφορικής τοπολογίας που αποβάλει. Έχουν ήδη εκφραστεί διάφορες τοποθετήσεις. Είναι σημαντικό λοιπόν η οδηγία αυτή να προχωρήσει και θα δούμε τελικά ποια είναι τα σημεία που θα ε, χρησιμοποιηθούν, θα περάσουν και θα χρησιμοποιηθούν ως μήνυμα περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε. Η κυρία Χάρκιν και μετά πάλι ο εισηγητής. Ευχαριστώ. Καταρχάς, έχω πολλούς Έχω όπως ε, και οι άλλοι ομιλητέ ε, να ευχαριστήσω τον κύριο Μπεναμιά για τις ε, προσπάθειές του. Είναι ένα δύσκολο θέμα ασφαλώ. Και κατάφερε να ξεύρει σε ένα μεγάλο βαθμό συμφωνία. Τον ευχαριστούμε λοιπόν για τη δουλειά του. Πολύ σύντομα θα υποστηρίξουμε τις συμβαστικές τοπολογίες ΑΒ και ΓΑΜΑ, ABC, την D διότι αναφέρεται σε αναθεώρηση της οδηγίας, η ε μας βρίσκει σύμφωνος, η 4, παράγραφος 4 είναι το κύριο ερωτηματικό και δεν έχουμε καταθέσει πολλές τροπολογίες εκ μέρους της ε, ομάδας μας. Θα δούμε τι είδους υποστήριξη σας ασφαλιστεί για την ε, παράγραφο αυτή αύριο. Και πάντως ευχαριστώ τον κύριο Μπεραμιάς για τη δουλειά του. Ευχαριστώ. Αν δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο, ο εισήγητης παρακαλώ. καλός για την 48. Ομολογώ ότι δεν ήμουν τόσο ενημέρωση. Αν μπορεί ξαδιβάζοντας την αλλάξω γνώμη, τι να πω, δεν βλέπω κανένα λόγο ιδιαίτερο. Κύριε Παλτασάρ. Μπαλτασάρη, προφορική ε, τροπολογία που έχετε καταθέσει εσείς νομίζω ότι ακολουθεί λίγο πολύ αυτά που είχε πει ο Επίτροπος Μπαρνιέ πρόσφατα. Συμβαστικά λοιπόν, συμβαστική τροπολογία νομίζω θα μπορούσε να είναι σχετικά ικανοποιητική σε σχέση με τα σχόλια τα οποία έχει να κάνει το Κοινοβούλιο για την οδηγία περί υπαρχής υπηρεσιών και τα προβλήματα που παρουσιάζει αυτή αλλά πέραν αυτού δεν μπορώ να πάω. Δηλαδή, με καλύπτει αρκετά η τροπολογία σας μεν, αποδεκτή μου φαίνεται ως συμβαστική μεν, πέραν αυτής όμως δεν μπορώ να προχωρήσω σε σχέση με τα σχόλια για την οδηγία περί ε, υπηρεσιών, ε, πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα σε σχέση με εκείνους που ωφελούνται ή ε, ζημιώνονται από την εν λόγω οδηγία. Και μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε και την ε, έκθεση επί της ουσίας ε, υπόψη αυτή τη στιγμή και ως εκ τούτου επιτροπή είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσουμε. Ξέρουμε για ποιους λόγους και τα λοιπά, έτσι είναι προσωπικοί λόγοι και σοβαροί λόγοι της ε, εισηγήτριας, αρμόδιας κατ' ουσίαν εισηγήτριας. Ε, μπορώ να σας προσεγγίσω κάπως, το, το έπραξα άλλωστε μόλις τώρα, αλλά πέραν αυτού δεν μπορώ να πω και ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρο. Αύριο το πρωί ψηφοφορία 9 και 30. Παρουσίαση μελέτη εφαρμογή των οδηγιών στο τομέα τη ασφάλεια και τη υγεία συνεργασία ω παράγον κόστου είναι το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Από την Marble Consorting έχουμε τον, την κυρία η οποία θα μας κάνει την παρουσίαση αυτή. Ε, αλλά θα ήθελα να δώσω το λόγο και στον κύριο Τάκλου από την ε, υπηρεσία του Μπιλμπάου για να μιλήσει μέχρι ότου έρθει η κυρία Βάου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να πω για την αρχική μου έκθεση, ε, εντύπωση πριν να διαβάσω την έκθεση, γιατί πρώτα έμαθα ότι έχει αναλυφθεί η διατύπωσή τη. Ήμουν κάπω επικριτικό πριν τη διαβάσω. Η εκτίση του Εμπέρ είναι πολύ γνωστή στου διάφορου κύκλου. Την έχουμε συζητήσει στην τρίμερη ε, διοικητική επιτροπή και στην Επιτροπή για την Οικία, την Ασφάλεια ε, και την Υγιεινή στον χώρο εργασία. Πλην ε, ενό όλα τα μέλη είχαν επικριτική στάση έναντι της ε, διαγραφής του όρου του μεσαίας επικινδυνότητας ε, ε, διαβαθμιζόμενου χώρου εργασίας. Έχουμε στην ίδια σύνδεση με τη Γενική Διεύθυνση για την Επιχειρηματικότητα και για την ιστορική αγορά. Έχω κάποια σχόλια λοιπόν αρχικά να κάνω για την έκθεση την οποία έχουμε μόλις δει. Βλέπουμε κάποια προβλήματα ως προς την έκθεση, επισήμανα ορισμένα από αυτά ήδη. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία ως προς τα οικονομικά ωφέλη της ε, ασφάλειας των χώρων εργασίας, αντίθετα από αυτά που ισχυρίζεται η έκθεση. Φερρυπίν, η ILO, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, ορίζει σε ποσοστό επί του ΑΕΠ 4% που απολένεται σε επίπεδο παγκόσμιο λόγω τέτοιων προβλημάτων και ταυτόχρονα ορίζει και με μια μελέτη της ε, τι είδους επιβάρυνση μπορεί να έχουν οι εργασιακές ε, ασθένειες που είναι 5% για τις βιομηχανικές χώρες όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αυστραλία πρόσφατα κατέγραψε με μια αρκετά εκτεταμένη ε, επίσημη έρευνα, κρατική έρευνα, ότι είναι 5,9 το ποσοστό απώλειας από το ΑΕΠ, ειδικά για την Αυστραλία, λόγω τέτοιου είδου ασθενειών. Και άλλη μια μελέτη από τη Φιλανδία καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η προώρη συνταξιοδότηση που σχετίζεται δηλαδή περί τα 57,6 έτη σταξιοδότηση αντί για τα 65 που ορίζεται ως νόμος προς συνταξιοδότηση μέχρι και 68 σήμερα πια. Ε, λοιπόν, η προώρη συνταξιοδότηση για λόγους υγείας ε, κοστίζει 25 δισεκατομμύρια στην Φινλανδία από το ΑΕΠ της. Σε προβολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε να κάνουμε με 2,5-3. Δηλαδή ποσό πενταπλάσιο αυτό της οικονομικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε στην ελληνική οικονομία. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό το χρόνο και κάθε χρόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, φρονώ ότι δεν αρκεί το να πούμε ότι 20.000 επιθεωρητές εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρκεί να επανεκπαιδευτούν για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Βεβαίως χρειάζεται βελτίωση αυτού του ζητήματος, αλλά και βελτίωση των όρων εργασίας. Έχουμε 25 με 27.000 άτομα με καθεστώς αναπηρίας και αναπηρική σύνταξη στην Ευρώπη και μόνιμες αναπηρίες που ε, αυξάνουν τον αριθμό των αναπήρων, των μόνιμων αναπήρων σε 2 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Έχουμε 20 εκατομμύρια ασθένειες ε, σχετικές με την ε, απασχόληση. Το Σουηδικό ε, Υπουργείο πρόσφατα εργασίας δηλώνει ότι 1,3, ένας στους τρεις εργαζόμενους βγαίνει από τον χώρο εργασίας για τέτοιους λόγους. Μεγάλη δαπάνη όπως καταλαβαίνετε. Κοστίζει πολύ αυτή η υπόθεση και έτσι από τα όσα βλέπω εδώ στη μελέτη διαπιστώνω ότι κανένας από αυτούς από τους οποίους ζητήθηκε συνέντευξη ε, δεν ήταν επιθεωρητής εργασίας, ούτε κάποιος ε, ε, επιχειρηματίας σε ειδική κατηγορία. 20.000 επιθεωρητές θα πρέπει να περάσουν αρκετό διάστημα πριν να αποδώσουν στις εργασίες, στην εργασία τους δηλαδή πριν να επισκεφθούν μία από τις μικρές ή μέσες επιχειρήσεις. Ε, υπολογίζεται μια επίσκεψη των δύο με τριών ωρών μία φορά το χρόνο για κάθε μικρομεσαία επιχείρηση της Ευρώπης με 20.000 επιθεωρητές εργασίας που έχουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν θα περάσει πολύ καιρό μέχρι να καταγράψουν τα φαινόμενα αυτά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, πέραν αυτών των ενισχυών όμως έχω και θετικά σχόλια για την έκθεση. Είναι καλή η παρουσίασή της. Από τα πορίσματα και τις συστάσεις της τα συμπεράσματά της τα περισσότερα είναι λογικά. Η επιστημονική δουλειά της υπηρεσίας μας αναγνωρίζεται ικανοποιητικά. Ο, το εργαλείο online, το διαδικτυακό εργαλείο, δηλαδή αξιολόγηση ε, εργασιακού κινδύνου αναγνωρίζεται ως σημαντικό και αποτελεσματικό και ύστερα από μια συνάντηση με τις Επιτροπές Μεακού. Ε, διαλόγου, κοινωνικού διαλόγου που συνάντησα σήμερα το πρωί και με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βλέπω ότι είναι αρκετά ικανοποιημένε από αυτό το εργαλείο αξιολόγηση του εργασιακού κινδύνου που έχουμε διαθέσει στο διαδίκτυο. Αυτή είναι η πρόταση που είχαμε εμείς προτείνει λοιπόν. Και για να ολοκληρώνω, βλέπω ότι πρόκειται για μια καλή έκθεση εν γέννη και θα ήθελα να ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αρκετά καλή αυτή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Σεβάστε λοιπόν από την Rambo Consulting για να μας κάνει την παρουσίασή της. Παρακαλώ, για την εφαρμογή της οδηγίας. Um, ευχαριστώ πολύ. Μόλις ήρθα. Ωραία. Φαίνεται στις οθόνες και η παρουσίασή μου understand Από ό,τι άκουσα, σχολιάστηκε κιόλα ε, η μελέτη μα. Άκουσα μόνο το τελευταίο τμήμα. Δεν φάνηκε να ήταν πολύ αρνητικό το σχόλιο. Είμαι εδώ για να σας παρουσιάσω την έκθεση αυτή σε σχέση με την εφαρμογή των οδηγιών ε, για την ασφάλεια και την υγεία στο ε, χώρο εργασίας ως παράγον κόστους τα, τους τελευταίους μήνες ε, εκπονήσαμε την μελέτη αυτή. Νομίζω πρέπει να βάλω τα γυαλιά μου. Ο στόχος λοιπόν ε, της ε, μελέτης είναι να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε καλύτερα τη σημασία της ε, επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας ε, ως παράγον ε, που συνεισφέρει ή μπορεί να συνεισφέρει στην οικονομική βιωσιμότητα των εταιριών, κυρίως των μικρομεσαίων. Επίσης, εξετάσαμε τις ενδεχόμενες συνέπειες των προτάσεων που υπευλήθησαν σε σχέση με την προσπάθεια μείωσης του διοικητικού φόρτου και ειδικότερα στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας ε, στο χώρο εργασίας. Επίσης εξετάσαμε σε ποιο βαθμό και πόσο καλά ε, πληρούνται αναλαμβάνονται οι υποχρεώσεις αυτές ε, κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επίσης εξετάσαμε κατά πόσο η μείωση των υποχρεώσεων ενημέρωσης ε, θα μπορούσε να είναι ένα εμπόδιο για την επίτευξη των ε, στόχων, των συνολικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την πρόληψη και την μείωση των ασθενειών και των ατυχημάτων που σχετίζονται με το χώρο εργασίας. Η μελέτη μας βασίζεται κυρίως ε, σε έρευνα ε, πολλών ε, εγγράφων που προέρχονται από τον Οργανισμό Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασία και όπως επίσης είχαμε και συμμετοχή πολλών εμπειρογνωμόνων και του οργανισμού που μόλις ανέφερα αλλά και κάποιων εργαζομένων. Λίγα λόγια για την ε, οργάνωση της ασφάλειας και της υγείας του χώρου εργασίας στην Ευρώπη. Βασική οδηγία 89-391 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ορίζει τις βασικές αρχές για την πρόληψη και την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων και επειδή είναι οδηγία πλαίσιο Υπάρχουν και πολλές άλλες οδηγίες που σχετίζονται. Νομίζω οι 19 και οι 20 ε, αφορούν πιο συγκεκριμένα ζητήματα ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας ε, Έγιναν και πολλές αναθεωρήσεις και η πιο πρόσφατη αναθεώρηση ήταν το 2004 όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπώνησε αναθεώρηση που έδειξε βασικές ε, αδυναμίες ε, στις ε, μικρές κυρίως επιχειρήσεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουν την νομοθεσία. Αφορούσε κυρίως, οι αδυναμίες αυτές αφορούσαν κυρίως τη συμμετοχή των εργαζομένων, την αξιολόγηση του κινδύνου, όπως επίσης και ε, με την κατάρτιση των εργαζομένων σε σχέση με ζητήματα ασφάλειας ε, και υγείας, όπως επίσης και ιδιαίτερα προβλήματα σε παραδοσιακούς ε, τομείς υψηλού κινδύνου, όπως οι οικοδομές και η γεωργία η μεταγραφή των ε, οδηγιών είχαν, ε, είχε οδηγήσει τα κράτη-μέλη να περάσουν από νομοθεσία που βασιζόταν κυρίως ε, σε μέτρα αποκατάστασης βλαβών σε πιο προληπτική προσέγγιση. Τώρα, οι βασικές αδυναμίες που εντοπίστηκαν προέρχονταν κυρίως από έλλειψη συγκεκριμένης και στοχευμένης ενημέρωσης σε τοπικό επίπεδο. Επίσης κακές υποδομές και έλλειψη δεξιοτήτων, έλλειψη γνώσεων σε σχέση με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία και όπως επίσης και έλλειψη λόγω της έλλειψης των πόρων ε, για την κατάρτιση του εργατικού δυναμικού αλλά και των διευθυντών. Όπως επίσης υπήρχε και πολύ κακή πρόσβαση σε αποτελεσματική και πιο εξειδικευμένη ε, τεχνική ενίσχυση. Κάποια από τα προβλήματα αυτά, κάποια από τα μειονεκτήματα αυτά αντιμετωπίστηκαν στο πλαίσιο τη Στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ασφάλεια και την Υγεία στον χώρο εργασία, που καλύπτει την περίοδο από το 2007 στο 2012 και ένα από του βασικού στόχου είναι 25% μείωση των ατυχημάτων στον χώρο εργασία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2012. Επίσης, για τη στρατηγική αυτή, η δράση σε κοινοτικό επίπεδο εστιάζεται κυρίως ε, στην ομοθεσία, την ενημέρωση και την απλοποίηση των μέτρων, ε, η καθοδήγηση και ανταλλαγή των πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, ενώ η περισσότερη συγκεκριμένη δράση λαμβάνεται από τους ενδιαφερομένους, ε, δηλαδή σε εθνικό επίπεδο. Τα εθνικά σχέδια δράσης δηλαδή είναι αυτά που πρέπει ουσιαστικά να ε, αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τις σχετικές αρχές ε, στο, ε, στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του διοικητικού φόρτου Αυτό θεωρείται ότι κατά κάποιο τρόπο αντίκειται στους ε, στόχους αυτούς ε, της ασφάλειας και της υγείας του χώρου Δηλαδή στον παρελθόν ε, υπήρχε ο στόχος της μείωσης 25% και υπάρχει ένα ακόμη ποσοστό 25% στο πρόγραμμα δράσης που αφορά τη μείωση του διοικητικού φόρου του. Ο στόχος είναι να μειωθεί κατά 25% και πάλι μέχρι το 2012. Φαίνεται ότι το 25% είναι ένα αρκετά δημοφιλές ποσοστό. Πρώτη φορά ε, εφαρμόστηκε το πρόγραμμα το 2009 με σκοπό να γίνει μια μέτρηση του διοικητικού φόρτου σε, πολλές, σε πολλούς τομείς πολιτικής και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανακοίνωση της Επιτροπής το 2009 που αναγνώρισε 13 ε, τομείς προτεραιότητας μεταξύ των οποίων είναι το περιβάλλον εργασίας και οι εργασιακές σχέσεις. Έξι συγκεκριμένες προτάσεις ε, για μέτρα μείωσης ε, υποβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τομέα του, περιβάλλοντος, του εργασιακού περιβάλλοντος. Δύο από τις προτάσεις αυτές έχουν ήδη εγκριθεί, ενώ έξι ε, ακόμη ε, είναι υπό, επεξεργασία και προσπαθήσαμε αυτές τις έξι που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί να τις εξετάσουμε περισσότερο στο πλαίσιο της μελέτης μας. Τώρα, όσον αφορά τι συγκεκριμένε προτάσει για την μείωση του διοικητικού φόρτου, η πρώτη πρόταση και η πιο διαφιλονικούμενη είναι η εξαίρεση πολύ μικρών ε, επιχειρήσεων, πολύ μικρών εταιριών ε, από, το, ε, από την εκπόνηση αξιολόγησης γραπτής, γραπτής αξιολόγησης των κινδύνων ασφάλειας και υγείας. Γιατί αφορά μία βασική υποχρέωση του κεκτημένου, συγκεκριμένα δηλαδή τη γραπτή αξιολόγηση. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι αυτό το συγκεκριμένο μέτρο θα τύχει ιδιαίτερη περιστατωμένη μελέτη από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόληση ε, πριν, ε, πριν, ε, πριν να ληφθεί οποιαδήποτε δράση στον τομέα αυτό. Επίση, ε, πρόκειται για μία από τις προτάσεις ε, για τις οποίες οι εμπειρογνώμονες ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο συμφώνησαν και αφορά, αφορά και τους εργαζομένους και, συγγνώμη, και εργοδότες ότι δεν είναι ο καλύτερος τρόπος δηλαδή να αντιμετωπιστεί το ζήτημα ε, υπήρχε συμφωνία σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι δεν πρέπει να απομακρυνθεί εντελώς η υποχρέωση της γραπτής αξιολόγησης για τις ε, ε, πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αντιθέτως προτείνεται μια προσέγγιση περισσότερο βασισμένη στον κίνδυνο ανάλογα με το είδος της εταιρείας και τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, μια πιο απλοποιημένη προσέγγιση δηλαδή. Οπότε, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι προκύπτει από τη δική μας τουλάχιστον μελέτη, ότι η διασυνοριακή άρση αυτής της υποχρέωσης ε, της γραπτής αξιολόγησης δεν είναι δυνατή ούτε για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει να ε, μελετηθεί περαιτέρω πριν από την τελική πρόταση. Η επόμενη πρόταση μείωσης μεταξύ των έξι που μελετήσαμε στο πλαίσιο της ε, μελέτης μας αφορούσε την διευκόλυνση ε, μεταγραφής των ε, της, της οδηγίας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων από τα κράτη-μέλη. Υπήρχε και πάλι ευρύτερη συνένεση στον τομέα αυτό ότι Πολύ καλή είναι η βελτίωση της κατανόησης ε, του στόχου της νομοθεσίας και του πώς μπορεί να εφαρμοστεί, όμως ε, υπάρχει, είναι ένας τομέας ε, που χρήζει μεγαλύτερης προσοχής. Δεν είναι δυνατό για μας, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, να πούμε τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό στις πραγματικές προσπάθειες πρόληψης των ατυχημάτων, για παράδειγμα, αλλά κατά πάσα πιθανότητα ο αντίκτυπος θα είναι μάλλον αρνητικός. Η επόμενη πρόταση μείωση ε, αφορά τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των επισκέψεων επιθεώρηση εργασία. Είναι κάτι το οποίο ακόμη εξετάζεται. Το να είναι πιο αποτελεσματικές οι επισκέψεις αυτές ε, με τη χρήση των πόρων, με την καλύτερη χρήση των εφισταμένων πόρων είναι κάτι που θεωρείται σε γενικές γραμμές ότι θα μειώσει το διοικητικό φόρτο και ότι δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ε, αρνητικών ε, συνεπειών. Βέβαια, το να είναι πιο αποτελεσματικές οι επισκέψεις εξαρτάται από το πόσο στοχευμένε θα είναι, να υπάρχει μια προσέγγιση που να εστιάζεται περισσότερο στον κίνδυνο, δηλαδή προς τις χώρες όπου υπάρχουν οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι και επίση να βρεθούν άλλοι τρόποι ε, αντιμετώπισης ε, των τομέων όπου οι κίνδυνοι δεν είναι τόσο μεγάλοι. Και υπάρχουν και κράτη-μέλη που θα μπορούσαν ε, να αποτελέσουν παράδειγμα ως προς, το ως προς τον τομέα αυτό των επισκέψεων της επιθεώρησης εργασίας. I have a bit of Συγγνώμη, αλλά είμαι κρυωμένη. Μία ακόμη πρόταση μείωση είναι η βελτίωση της καθοδήγησης ε, για τις ε, εταιρείες ε, του κατασκευαστικού τομέα, για τις ε, οικοδομές των εργοταξίων. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το θέμα αυτό. Δεν υπάρχουν δηλαδή αρνητικές συνέπειε ε, ως προς την βελτίωση αυτής της καθοδήγησης ε, για τον κατασκευαστικό τομέα. Επόμενη πρόταση αφορά τους ε, κινδύνους αξιολόγησης ε, Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια και την Υγεία ε, στο χώρο εργασίας αναπτύσσει ένα εργαλείο το οποίο μάλλον κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση γιατί είναι αρκετά διαδραστικό, βοηθά την αξιολόγηση κινδύνου και ειδικότερα από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γενικά θεωρείται κάτι πολύ θετικό, μια πολύ θετική ε, εξέλιξη. Τα μόνα ζητήματα που προέκυψαν είναι πόσο προσαρμοσμένη θα είναι η προσέγγιση αυτή στους διάφορους τομείς και στα διάφορα είδη επιχειρήσεων και ο βαθμός ακριβώς της προσαρμογής ε, είναι πάρα πολύ σημαντικός προκειμένου να είναι χρήσιμα τα εργαλεία που αναπτύσσονται. Πρέπει λοιπόν ε, το εργαλείο αυτό να προσαρμοστεί πάρα πολύ καλά στις ιδιαίτερες ανησυχίες ε, πολύ συγκεκριμένων ε, επιχειρήσεων. Και η τελική πρόταση μείωσης ε, διοικητικού φόρτου αφορά τη βελτίωση τρόπων ε, επεξεργασίας βασικών πληροφοριών για τους ε, καρκινογενείς παράγοντες και αυτό δεν είναι εύκολο να εξεταστεί γιατί υπάρχει αναθεώρηση αυτή τη στιγμή της οδηγίας και επομένως σε αυτό το στάδιο είναι αδύνατον να διαπιστώσει κανείς ποιες θα είναι οι συνέπειες η διαπίστωση αυτή μπορεί να γίνει μόνο αυτή τη στιγμή ε, αναθεωρηθεί η οδηγία και έχουμε τις νέες ε, προτάσεις υπόψη μας. Αυτές λοιπόν ε, ήταν οι έξι προτάσεις που ακόμη δεν έχουν εγκριθεί και τις οποίες είχε υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι περισσότερες από αυτές τις προτάσεις, και νομίζω ότι είναι σαφές από όλα όσα είπα, ε, δεν δημιουργούν προβλήματα, κυρίως ε, με την εξαίρεση της πρώτης όμως, ε, όσον αφορά την άρση των υποχρεώσεων γραπτής αξιολόγησης κινδύνου από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αυτή είναι η μόνη πρόταση η οποία, από την οποία προέκυψαν κάποια αρνητικά σχόλια. Κάτι ακόμη που θελήσαμε να εξετάσουμε είναι αν μπορούμε να καταδείξουμε σαφέστερα την συμμόρφωση με τους ε, κανόνες για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας. θα έλεγε κανείς ε, ότι όντως ε, είναι σημαντικό να γίνει κάτι τέτοιο, ότι έχει κάποιο όφελος, όμως πολλές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταδείξει κανείς την άμεση σχέση μεταξύ των δύο, γιατί δεν υπάρχουν και πολλά ε, στοιχεία στον τομέα αυτό. Υπάρχουν κάποιες άμεσες συνέπειες οι οποίες είναι ορατές, μπορούν εύκολα να ε, προσμετρηθούν, όπως για παράδειγμα η μείωση του κόστους ε, που ε, έχει να κάνει με τη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων ή των ασθενειών, σημαίνει λιγότερες άδειες μεταποδοχών, σημαίνει λιγότερη, αποχή, λιγότερη απουσία των εργαζομένων από τη δουλειά τους, σημαίνει επίσης μείωση των ετοιμάτων αποζημίωσης. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι απολύτως σαφή, είναι κάτι το οποίο μπορούν ε, να κατανοήσουν οι περισσότερες εταιρείες. Υπάρχουν επίσης και οικονομικά ωφέλη με την, ε, από τη συμμόρφωση με τους ε, κανόνες για την ασφάλεια και την υγεία. Στο χώρο εργασίας όμως υπάρχουν και κάποια πιο έμεσα αποτελέσματα, κάποιες πιο έμεσες συνέπειες που χρήζουν περαιτέρω μελέτης. Γιατί ο παραδοσιακός τρόπος εξέταση των άμεσων συνεπειών μπορεί να μην επαρκεί. Είναι σημαντικό να ε, δούμε και την πτυχή των ε, μη απτών. Είναι ζητήματα δηλαδή τα οποία, μη των μη απτών συνεπειών, είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με τόσο από τα πράγματα όπως η μείωση του κόστους για παράδειγμα και αυτό έχει να κάνει με την καλύτερη φήμη της εταιρεία, όλο και περισσότερο είναι σημαντικό για τους καταναλωτές σήμερα να αγοράζουν ε, αγαθά και υπηρεσίες από εταιρείες ε, που ε, τους αντιμετωπίζουν με τον σωστό τρόπο. Επομένω, η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και μπορεί να είναι ένα έμεσο όφελος από την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στον χώρο εργασίας σε μια εταιρεία. Η βελτίωση της οργάνωσης της εργασίας πολλές φορές ε, υπάρχουν κίνδυνοι που προκύπτουν από κακώς προγραμματισμένη ή κακώς συντονισμένη εργασία. Η βελτίωση της οργάνωσης ε, και του συντονισμού ε, των εργασιών μιας επιχείρησης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα πιο αποτελεσματική εργασία αλλά και μείωση των κινδύνων. Ένα καλό εργασιακό περιβάλλον και επομένως αυξημένη ικανοποίηση των εργαζομένων είναι επίσης ένα μάλλον έμεσο ε, μια άμεση, ε, ε, συγγνώμη, έμεση συνέπεια ενός βελτιωμένου εργασιακού περιβάλλοντος που σέβεται περισσότερο τους κανόνες ασφάλειας και υγείας. Να σα πω και ορισμένα παραδείγματα. Ανέφερα προηγουμένως ε, την βελτίωση τη οργάνωσης και του συντονισμού του χώρου εργασίας. Ε, υπήρξαν πολλά παραδείγματα, όπως ε, για παράδειγμα η ροή εργασιών σε εργοτάξια, για παράδειγμα, που συνεργάζονται πολλές εταιρείε και είναι πολύ εύκολο να μπουν ο ένας στα χωράφια του άλλου και επομένως τα πράγματα μερικές φορές είναι δύσκολα και καθυστερεί η υλοποίηση του έργου. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα παράδειγμα ε, διπλού ωφέλους, ε, βελτίωσης του χώρου εργασίας και βελτίωσης της παραγωγικότητας. Ένα ακόμη παράδειγμα είναι η καλύτερη ε, εργονομία στις εταιρείες, κάτι το οποίο έχει ως αποτέλεσμα ότι ε, ένας άνθρωπος που χρησιμοποιεί το ποντίκι του υπολογιστή του πονάει λιγότερο στην πλάτη για παράδειγμα και αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την παραγωγικότητά του, την αποτελεσματικότητά του. Και ένα τρίτο παράδειγμα είναι κάτι που ανέφερα προηγουμένως και αφορά την ε, κοινωνική εταιρική ευθύνη για τους υπεργολάβους και για τους ε, παροχής υπηρεσιών που πρέπει επίσης να βελτιώσουν ε, τις προδιαγραφές τους ε, για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας. Τέλος, σε σχέση με το οικονομικό όφελος, είναι το κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο σε κάθε κράτος μέλος ε, διαφέρει. Και σας δίνουμε και ένα παράδειγμα στη μελέτη μας. Υπάρχουν διαφορές στις υποχρεώσεις των ε, κρατών ε, μελών για την πληρωμή, την αμοιβή των εργαζομένων που έχουν πάρει άδεια, για παράδειγμα. Υπάρχουν σοβαρές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Στις κάτω χώρες, για παράδειγμα, Δύο χρόνια μπορούν να πάρουν ε, ε, άδεια μεταποδοχών ε, οι εργαζόμενοι. Στη Γερμανία 42 μέρες είναι η αντίστοιχη περίοδος, η Ουγγαρία είναι 15 ημέρες και η Ιρλανδία δεν υπάρχει νομική υποχρέωση ε, άδειας μεταποδοχών προς τους εργαζομένους. Υπάρχουν λοιπόν τεράστιες διαφορές και γι' αυτό το λόγο Υπάρχουν και πάρα πολύ μεγάλες διαφορές ε, στα κίνητρα των εταιριών ε, για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στον χώρο εργασίας και είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν και άλλα πολλά παραδείγματα διαφορών μεταξύ των κρατών μελών και είναι κάτι το οποίο πρέπει να ληφθεί και αυτό υπόψη όταν προσπαθούμε να πείσουμε τις χώρες για το οικονομικό όφελος ε, της βελτίωσης των προδιαγραφών ε, ασφάλειας και υγείας. Then moving on to um, SMEs and, um, <clears throat> and their uh, compliance with obligations. Παίρνουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και την τήρηση από πλευρά του των υποχρεώσεων περί υγείας και ασφάλεια του χώρου εργασία. Βεβαίω, σημειώνουμε ότι το μέγεθος μια επιχειρήση είναι πολύ σημαντικό για το βαθμό στον οποίο θα τηρήσουν την νομοθεσία και τις προδιαγραφές της. μικρότερε επιχειρήσει. είναι πολύ πιο πιθανό να μην έχουν το σύστημα καταγραφής και διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας που απαιτείται. Επίσης, φραγμή σχετική με την γνώση της κατάστασης, δηλαδή έλλειψη συνειδητοποίησης, γνώση, ενημέρωσης για τους ε, κανόνες αυτούς, η έλλειψη γνώσεων ως προς την, τις συνθήκες ασφαλείας, προστασίας ε, της ε, υγείας και υγιεινής, είναι παράγοντες οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ε, προσπάθεια να ενισχυθεί το επίπεδο υγεία, ασφάλεια και υγιεινή στον χώρο εργασία. Στην επόμενη διαφάνεια δεν ξέρω αν βλέπετε τι λεπτομέρειε. Πάλι έχουμε αριθμητικά στοιχεία τα οποία προέρχονται από κάποιε πηγέ δικέ μα και που δείχνουν ε, ικανοποιητικά πιστεύω την κατάσταση. Έχουμε εδώ στα διάφορα χρώματα το μέγεθος της επιχείρησης Μικρότερε επιχειρήσει είναι αυτέ που έχουν το σκούρο χρώμα, οι μεγαλύτερε αυτέ που έχουν το πιο ανοιχτό χρώμα. Οι δύο πρώτες σας στήλε ασχολούνται με την ύπαρξη, εφόσον υπάρχει βέβαια ε, οργάνωση, και η δεύτερη με την αξιολόγηση. Βλέπετε με μεγάλη απόκληση μεταξύ των δύο κατηγοριών επιχειρήσεων. Οι μικρότερες δηλαδή επιχειρήσεις κυρίως αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες στην υπόθεση αυτή. Τι μπορεί να γίνει τώρα για να βελτιωθεί το επίπεδο της υγείας και ασφάλειας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. από τις μελέτες μας βλέπουμε ότι δεν είναι η καλύτερη λύση το να μειωθούν οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις. Μάλλον θα ήταν σκοπιμότερο να προσαρμοστούν ανάλογα με το τύπο της επιχείρησης οι υποχρεώσεις που τους εμπίπτουν και πάλι με προσεγγίσεις επικινδυνότητας ή αξιολόγηση κινδύνου που ε, εστιάζονται ακριβώ στα σημεία στα οποία ανάλογα με τον τομέα ή το είδο τη επιχείρηση είναι υψηλότερο το ποσό του κινδύνου και απλουστευμένε διαδικασίε που βελτιώνουν τα συστήματα Φιρπή είναι ένα σύστημα online που θα μπορούσε να βοηθήσει τις μικρότερες επιχειρήσεις ώστε να αντεπεξέλθουν στις ε, υποχρεώσεις τους. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι η δουλειά που έχει γίνει και που συνεχίζεται. Και εδώ αναφέρομαι στα όσα έχουμε εμείς μπορέσει να κάνουμε βάσει τους δικούς μας ε, πόρους. Όταν έχουμε να κάνουμε μικρότερες επιχειρήσεις, ε, η επικοινωνία ένας προς έναν, ε, ενώπιος ενωπίο λίγο πολύ, είναι πολύ πιο αποτελεσματική από ε, προσπάθειες επικοινωνιακές ή ενημέρωσης μεγάλης κλίμακας. Μέσα από τις επιχειρήσεις με τις οποίες ή τις οργανώσεις με τις οποίες συνεργάζεται μια τέτοια επιχείρηση, την τράπεζα ή την ασφαλιστική, την υπηρεσία, την ε, ασφαλιστική εταιρεία με την οποία έχει συνεργασία, μπορούμε νομίζω να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα και ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε μια προσέγγιση είτε εθνικού χαρακτήρα είτε τομεακού συμπληρωματικά ώστε να ε, υπογραμμίζονται τα πλεονεκτήματα της ε, τήρησης των υποχρεώσεων στον τομέα αυτών. Κλείνω αναφερόμενοι αναφέροντας τους ε, αναδιόμενους κινδύνους, το νέο τομέα, δηλαδή τους νέους κινδύνους και ιδιότερα, ιδιαίτερα τις τρεις κύριες ομάδες ή κατηγορίες αναδειωμένων κινδύνων ως προς την υγεία και ασφάλεια, μειοσκελετικές ε, διαταραχές, μη σίγμα δέλτα δηλαδή, MSD στα αγγλικά, που είναι γνωστές πιστεύω, οι ψυχοκοινωνικές διαταραχές ή προβλήματα όπως το στρες κτλ. Και, και τομεί που έχουν να κάνουν, ε, τομέα μάλλον κινδύνου που έχει να κάνει είτε με, το, ε, με την παρουσία επικίνδυνων ουσιών, νέων τεχνολογιών και άλλα στοιχεία ή ε, ζητήματα που έχουν να κάνουν με σωματικό κίνδυνο. Επίσης, η ζητηματα που εχουν να κανουν με σωματικο κινδυνο Επίση, η καταπολεμηση των ε, ατυχημάτων στον χώρο εργασία μια εκστατεία που είχε γίνει και που βλέπουμε ότι έχει αποδώσει, οδήγησε σε μείωση των ατυχημάτων στον χώρο εργασία, με ταυτόχρονη όμω αύξηση των προβλημάτων υγείας και των εργασιακών ασθενειών, επαγγελματικών ασθενειών. Σαν να έχει μετακυλήσει το πρόβλημα από το εργατικό ατύχημα στην εργασιακή πάθηση ή νόσο. Και πάλι, όπως είπε, υπάρχουν και οι τρεις νέες κατηγορίες κινδύνων που εμφανίζονται τώρα, που επιβαρύνουν την κατάσταση. Στις ε, μειοσκελετικές διαταραχές έχουμε να κάνουμε εδώ με το πιο συνηθισμένο φαινόμενο ε, προβλημάτων υγείας, που σχετίζονται με το χώρο εργασίας, είναι το τα δύο τρίτα των προβλημάτων υγείας και το δεύτερο συνηθέστερο είναι αυτό των ψυχοκοινωνικών διαταραχών που σχετίζονται συχνά με τις τρεις συνθήκες εργασίας ή απασχόλησης μέσα στον νέο κόσμο τον οποίο έχουμε αντιμετωπίσουμε. Ο εργαζόμενος έχει νέες συμβάσει με διαφορετικούς όρους, με μεγαλύτερη ανασφάλεια, ε, με μικρότερη ασφάλεια μάλλον προς την θέση εργασίας. Έχουμε περισσότερη ε, περισσότερο ηλικιωμένο πληθυσμό, πιο κατακαιρματισμένη ε, κατακαιρματισμένο εργατικό δυναμικό με ομάδες διαφορετικές όπως γυναίκες, ηλικιωμένων κτλ. που σημαίνει ότι, υπάρχουν, ε, ότι έχουμε διαφορετικά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε ανάλογα με την κατηγορία των εργαζομένων. Έχουμε περισσότερη ένταση εργασίας και αυτό έχει να κάνει βέβαια με την ισορροπία ε, της εργασίας με τον ιδιωτικό βίο. Η εντατικοποίηση της ε, τεχνολογίας ε, στην ζωή μας έχει, να, έχει σαν συνέπεια ότι χάνεται η διάκριση μεταξύ απασχόλησης, η εργασίας και του ιδιωτικού βίου. Και επίσης έχουμε πολύ υψηλή συναισθηματική επιβάρυνση στον χώρο εργασίας, δηλαδή δεν υπάρχει η διαπροσωπική σχέση. άλλοι αναβιώμενοι κίνδυνοι. Δεν θα αυτέ στι λεπτομέρειε, αλλά έχουμε να κάνουμε τι νανοτεχνολογίε, του βιολογικού κινδύνου. Με περιορισμένη γνώση των επιπτώσεών του, ιδιαίτερα όσον αφορά την νανοτεχνολογία, πράγμα που έχει σαν συνέπεια να μην είναι δυνατόν και να εντοπιστεί ή να αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά ο κίνδυνος που προέρχεται από αυτές τις νέες τεχνολογίες, νανοτεχνολογίες. Άρα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή να αποδοθεί σε αυτό. Ιδιαίτερα τα επόμενα χρόνια. για τους ε, νέους αναδυόμενους ή ενισχυόμενους παράγοντες κινδύνου. Οι μειοσκελετικές διαταραχές Φερρυπίν δεν είναι καινούριο κίνδυνος αυτός, καθε, ε, αυτός καθεαυτός, αλλά έχει ενισχυθεί ιδιαίτερος η ενισχυομενους παραγοντες κινδυνου οι μειοσκελετικες διαταραχες φερρυπιν δεν ειναι καινουριο κινδυνος αυτος καθεαυτος αλλα εχει ενισχυθει ιδιαιτερο η παρουσια του και ίσως έχει και περισσότερη ε, προσοχή προσελκύσει, δηλαδή ο εργαζόμενος είναι λιγότερο διατεθειμένος να υποφέρει από μια μειοσκελετική διαταραχή και αντιδρά περισσότερους, γι' αυτό εμφανίζεται σε πρώτη θέση επικαιρότητα. Η νομοθεσία ε, και ο προσανατολισμός τους προς την ε, πρόληψη μας οδηγεί στο εξής συμπέρασμα. Οι κίνδυνοι σε μεγάλο βαθμό φαίνεται να καλύπτονται από την υφιστάμενη οδηγία, δηλαδή κενό νομοθετικό, ανάγκη για νέο νομοθέτημα δεν φαίνεται να υπάρχει. Ίσως σε, νέο, σε κάποιους τομείς όπως η νανοτεχνολογία να χρειάζονται πιο ειδικέ ε, δράσεις, αλλά γενικά η νομοθεσία καλύπτει τους κινδύνους εν γέννη. Πλην όμως υπάρχει ανάγκη να εξεταστεί περισσότερο το λειτουργικό επίπεδο έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν χρειάζονται νέα εφαρμοστικά μέτρα ή χρειάζεται να δοθεί περισσότερη προσοχή στα εφαρμοστικά μέτρα. Το περιβάλλον επίσης αλλάζει συνέχεια και να χρειάζεται μια ε, ιδιαίτερη εστίαση, προσαρμογή και προσαρμοστικότητα. Συμπληρώνω επίση ότι χρειάζεται να αντιμετωπιστούν και οι φυστάμενοι, αλλά και οι νέοι κίνδυνοι παλαιοί. Οι φυστάμενοι δηλαδή κίνδυνοι δεν εξαφανίζονται αυτόματα, παραμένουν, υπάρχουν ακόμα δηλαδή κίνδυνοι των εργασιακών ατυχημάτων, των εργατικών ατυχημάτων ή τα παραδοσιακά προβλήματα υγεία που σχετίζονται με την εργασία. Άρα δεν πρέπει να τα λησμονούμε και αυτά ενώ ταυτόχρονα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και στους νέους κινδύνους που εμφανίζονται. Ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο είναι το σχετικό με τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. Πολλοί είναι αυτοί οι εκπρόσωποι με τους οποίους μιλήσαμε που λένε ότι είναι οι πιο ε, δυσδιάκριτοι κίνδυνοι, είναι αυτοί που είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπίσει κιόλας κανείς, έχουν να κάνουν με τον τρόπο με το χαρακτήρα, με τον τρόπο εργασίας δεν είναι κάτι δηλαδή, το αντικειμενικά προσδιοριζόμενο και είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν ως εκ τούτου και χρειάζονται νέα μέσα και κατευθυντήριες γραμμές. Καταλήγω τώρα με τις, με, με τις συστάσεις μας. Ήδη το έχουμε αναφέρει αρκετές φορές. Υπάρχει μια ανάγκη να εισεχθούν προσεγγίσεις στηριζόμενες στον κίνδυνο ή προσαρμοσμένες περισσότερο στους ιδιαίτερους κινδύνους που χαρακτηρίζουν κάποιους τομείς, ε, τύπους εταιριών, και ενδεχομένω σε συνδυασμό με απλουστευμένε διαδικασίε για τι μικρότερε επιχειρήσει. Αυτό είναι προτιμότερο από το να ε, απαλληφθούν οι προποθέσει για τι μικρότερε επιχειρήσει. Επίση είναι σαφέ και ίσω είναι το σαφέστερο πώς προκύπτουν από την μελέτη μας, γιατί μας ζητήθηκε να εξετάσουμε ποια είναι τα ωφέλη, οικονομικά ωφέλη των συνθήκων υγεία υγιεινής και ασφάλεια του χώρο Ναι, ε, ασφαλώ δεν υπάρχουν ε, απτά στοιχεία ωφέλους, άρα ίσως εάν πιστούν οι επιχειρήσεις ότι το να τηρούν ε, εάν στόχος μας είναι να πιστούν οι επιχειρήσεις το να τηρούν ε, τις προδιαγραφές ε, τις συμφέρει, τότε χρειαζόμαστε πολύ πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Στοιχεία τα οποία να μπορούν, με τα οποία να μπορούν να ταυτιστούν, στα οποία να μπορούν να δουν άμεσο συμφέρον. Αυτά βέβαια θα πρέπει να εξασφαλιστούν χάρη σε μια έρευνα. Και επίσης σχετικό με αυτό βλέπουμε ότι οι μικρές ε, επιχειρήσεις θα πρέπει να ενθαρρύνονται στην καλύτερη παρακολούθηση των οικονομικών τους επιδόσεων στο τομέα της ε, υγείας, ασφάλειας και υγιεινής στον χώρο εργασίας. Αν το καταφέρουμε αυτό ασφαλώς θα είναι πιο εύκολο να αναλάβουν και το διοικητικό βάρος. Επίσης είναι σημαντικό να δούμε τις διαφορές μεταξύ των εθνικών δεδομένων δομών. Ένα παράδειγμα ήταν η περίοδος κατά την οποία μια επιχείρηση καλείται να καταβάλει επίδομα ή μάλλον να καταβάλει μισθό κατά την περίοδο της ε, ε, άδειας για λόγους ασθενείας του προσωπικού της. Άρα εδώ χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο περισσότερες προσαρμογές σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο κοινωνικών εταίρων, παραγόντων που εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή και βέβαια των εθνικών αρχών που έχουν τις σχετικές αρμοδιότητες. Επίσης, η σύστασή μας είναι στο βαθμό του δηλαδή όταν γίνονται οι εκστρατείες ενημέρωσης να υπάρχει απευθείας επικοινωνία και άλλη λεπίδραση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλίσουμε καλά αποτελέσματα. Εν τέλει, χρειάζεται και να συμπληρωθούν τα παραδοσιακά εργαλεία που έχουμε στη θέση μας, την υπόθεση αυτή, με εργαλεία τα οποία να μπορούν να εντοπίσουν τους νέους και αναδυόμενους κινδύνους, όπως με τις νέες τεχνολογίες και ο τρόπος ενημέρωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα έχει μεγάλη σημασία, η επικοινωνία δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή ήταν η παρουσίασή μου. Καλύπτει αρκετά, πιστεύω, αρκετούς τομείς, ποικίλου τομείς. Ελπίζω όμως να διαφαίνεται ο μύτος της Αριάδνης που μας καθοδήγησε σε αυτό το κείμενο, σε αυτή την παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ. Για την παρουσίασή σας, ο λόγος που ακούσαμε τον προηγούμενο μελητή από εσάς ήταν ότι ξεκινήσαμε λίγο νωρίτερα. αυτό ήταν ο λόγος, μην ανησυχείτε. Είχαμε μια επισκόπηση τη όλη σα δουλειά πριν την παρουσιάσετε εσεί οι ίδια. Καταλαβαίνω ότι σα παραξένεψε κάπω, κανονικά όμω δεν θα είχε συμβεί. Έχω δύο ομιλητέ αυτή τη στιγμή και αρκετέ παρατηρήσει από μένα την ίδια. Η κυρία Μωράν Σαρτιέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βρισκόμαστε τώρα σε ένα θέμα, υγεία και ασφάλεια στην εργασία, που μας κινητοποιεί πλήρως. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το να δούμε τον αντίκτυπο στο κόστος για τις επιχειρήσεις είναι ένας τρόπος να αντιλαμβάνεται κανείς τα πράγματα. Όμως, ίσως να μην είναι η κεντρική πύλη εισόδου στην ουσία του θέματος. Αυτό που μας ε, συγκινεί τους μεν και τους δε είναι η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στις θέσεις εργασίας τους. Ε, αυτό πρέπει να είναι η πρώτη μας μέρημνα. Ε, το οικονομικό όφελος για την επιχείρηση έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Μετά τον στόχο τον ανθρώπινο, τους ανθρώπους δηλαδή. Αυτό είναι που μας ε, αφορά πάνω απ' όλα. Η παρουσίαση αυτής της παρουσίασης βέβαια με τόσες λεπτομέρειες μας δίνει μια νέα πρόπτικη για το όλο θέμα. Γι' αυτό θα ήθελα να θέσω κάποιες ερωτήσεις μετά από την παρουσίαση αυτή που κάνατε γιατί θα είχα θα ήθελα κάποιε συγκεκριμένε λεπτομέρειε. Πρώτα απ' όλα, μας είπατε ότι υπάρχουν 20 εκατομμύρια μικρομεσαίε επιχειρήσεις, 20.000 επιθεωρητές, δεν τον αριθμοί κατά προσέγγιση, σχεδόν ακριβής, αυτό είπατε. Μπορούμε να έχουμε πολλές απαιτήσει από τον έλεγχο, την επιθεώρηση ή μπορούμε να φανταστούμε ότι η επιθεώρηση θα είναι θετική. Πρέπει δηλαδή η επιθεώρηση να συμπληρώνεται με κυρώσεις ή και σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός μειώνει σοβαρά την σημασία του όλου ζητήματος. Μήπως μπορούμε να φανταστούμε λοιπόν ότι είναι άλλος ο ρόλος των επιθεωρητών, πιο επικοδομητικός για την επιχείρηση ώστε να γίνουν και οι ίδιοι φορείς της εξέλιξης για την επιχείρηση με ενεργό συμμετοχή. Ποια είναι η δική σας η αντίληψη της ε, επιθεώρησης και των επιθεωρητών. Έπειτα, με τη γραφική παράσταση που μας δείξατε, είδαμε ότι η διαφορά στο μέγεθος των επιχειρήσεων έχει σοβαρό αντίκτυπο στο πώς αντιμετωπίζετε το θέμα της υγείας και ασφάλειας στην επιχείρηση. Θα μπορούσατε να μας δώσετε αναμέγεθος επιχείρησης και ανα κλάδο επιχειρηματικό το τι προσαρμογές ε, γίνονται στην πράξη ή θα μπορούσαν να γίνουν στην πράξη προκειμένου να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες. Δεν μπορούμε να ζητούμε το ίδιο και με τον ίδιο τρόπο από επιχειρήσεις ε, στον τομέα της γεωργίας λόγου χάρη, μας είπατε ότι είναι ένας τομέας όπου υπάρχουν πολλά εργασία κατοχήματα ή μάλλον όπου γνωρίζουμε ότι μπορεί να μιλάμε εδώ για επιχείρηση 30 ατόμων. Δεν μπορούμε λοιπόν να ζητάμε τα ίδια με αυτή την επιχείρηση όπως με μια άλλη που έχει πολύ άριθμο εργατικό προσωπικό. Το συσχετισμό λοιπόν με τους κλάδους και το μέγεθος θα θέλαμε. Τρίτη παρατήρηση. Έχετε βρει το συσχετισμό μεταξύ των παθολογιών, των ψυχοπαθολογιών που λέτε ότι βρίσκονται σε αύξηση της επιχειρήσης και το επίπεδο κοινωνικού διαλόγου στις επιχειρήσεις αυτές. Διότι εκεί θα μπορούσαμε να βρούμε προσεγγίσεις τελείως καινούργιες, ιδίως για τις μικρές επιχειρήσεις, όπου ξέρουμε ότι η εγκύτητα και ο κοινωνικός διάλογος είναι πολύ καθοριστικές. Μπορεί να οργανώνονται τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο όπω στι μεγάλες επιχειρήσεις άραγε. Και δύο τελευταίε ερωτήσει που ήθελα να σα κάνω. Η από απόσταση εργασία, εκεί θα θέλαμε να αρχίσουμε να έχουμε κάποιες πρώτες ιδέες να ξέρουμε τι γίνεται με την παρακολούθηση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων που εργάζονται από απόσταση. Είναι δύσκολο αυτό από ψυχολογικής και μόνο άποψης, διότι υπάρχουν προβλήματα απομόνωσης. Και έπειτα την ε, εργασία αυτή την ε, προορίζουμε μόνο για ανθρώπους που δεν έχουν πολύ καλή κατάσταση υγείας σε ορισμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων. Υπάρχει αυτό εναλλακτική, υπάρχουν άλλε εναλλακτικέ, πώ το βλέπετε. Και δεύτερη ερώτηση, τελευταία θέλω να σα κάνω. Πώ βλέπετε εσεί, μέσω τη μελέτη που κάνατε, του μισθωτού που έχουν μακρές, μακρά, παθολογικά προβλήματα με συμπτώματα που επαναλαμβάνονται να κυκλώνονται, όπως ε, καρκίνους οι εργαζόμενοι και για την ψυχολογική τους υγεία να καλό να επιστρέφουν στην εργασία τους. Πώς μπορεί λοιπόν αυτό να αναλαμβάνεται ως ευθύνη από την επιχείρηση, αυτές οι πολύ συγκεκριμένε περιπτώσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκρίνα και μετά ο κύριος Κρίστανσον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήδη ο τίτλος μου, με προβλημάτισε λίγο, διότι μιλάμε για τον παράγοντα του κόστους. Για μένα η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία είναι επένδυση. Επένδυση που γίνεται προ όφελο των ίδιων των επιχειρήσεων. Όταν λοιπόν μιλάμε για μείωση του διοικητικού φόρτου, εμένα αυτό μάλλον με σοκάρει. Διότι νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μειώσουμε αισθητά σε κάποιου τομεί το κόστο και όχι στην υγεία και την ασφάλεια. Εδώ πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι είναι σημαντικότατο σήμερα παντού στην Ευρώπη, όπου γίνεται λόγος για την ε, επιμήκυνση του χρόνου εργασίας των ανθρώπων. Ε, εδώ λοιπόν η υγεία και η ασφάλεια είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει και σε σχέση με τους ε, πιο ηλικιωμένους πολίτες. Πώς θα παραμένουν στην τομέα της απασχόλησης, ιδίως αν είναι μάλιστα επώδυνη η εργασία τους. Νομίζω λοιπόν ότι και αυτό το ζήτημα είναι σημαντικό. Θα πρέπει να το δούμε και από την ε, πρόπτικη της υγείας στην εργασία. Τώρα για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση των κινδύνων στις ιδιαίτερα μικρές επιχειρήσεις. Εδώ προφανώς δεν συμφωνώ καθόλου. Ακόμη και αν λέγεται ότι απλώ δεν θα χρειάζεται η γραπτή αξιολόγηση. Δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει αξιολόγηση αν δεν γίνει γραπτός η εργασία αυτή η γραπτή θα αξιολογείται κάθε 6 μήνες, κάθε χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει έστω ένα έγγραφο, ένα χαρτί. Δεν μπορούμε να άρουμε αυτήν την ε, υποχρέωση αξιολόγησης και εγώ μπορώ να σας πω στην πράξη, επειδή υπήρξα διευθύντρια ανθρωπινοδυναμικού δυναμικού σε μια μικρή σχετικά επιχείρηση, μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι είτε είναι μεγάλη είτε είναι μικρή επιχείρηση, όλα είναι αποφασιστική σημασίας όταν δεν μπορεί να επειδή είσαι εργαζόμενο σε μια μικρή επιχείρηση με τρία άτομα να ασχολούνται ε, ο εργοδότη λιγότερο με την υγεία και την ασφάλειά σου. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, κυρίω γιατί σε πολλού τομεί έχουν γίνει σημαντικά βήματα πρόοδου ω προ την υγεία και την ασφάλεια. Και επειδή υπήρξε μια σοβαρή βελτίωση τη παραγωγικότητα των επιχειρήσεων που έκαναν αυτέ τι επενδύσει. Είναι λοιπόν επένδυση, σα λέω πάνω απ' όλα. Όσο για το σκέλο τη ε, θα συμφωνήσω εδώ με την συνάδελφο, με την Μπέκ. Διότι προτιμώ την πρόληψη παρά την αστυνόμευση, είναι πάντα το καλύτερο. Αλλά αυτό είναι σαφώ θέμα προτεραιότητα και κάτι που μου φάνηκε κάπω παράξενο για τις επιχειρήσεις και το καλό όνομα που έχουν σε σχέση με την ε, ε, υγεία και την ασφάλεια για τους διαγωνισμού σαφώς θα μπορούσε να τους δίνεται το προβάδισμα όταν τα πάνε καλύτερα και στο περιβάλλον και στην υγεία και την ασφάλεια. Όμως, σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις που ο πελάτης τους είναι ο μεμονωμένος καταναλωτής, Πολλέ φορέ αυτό είναι το θέμα και τη. Εκεί παίζει ρόλο και το κόστο. Δηλαδή, αν κοστίζει ακριβότερα για τι επιχειρήσει αυτέ, ε, θα είναι και περιορισμένε προσπαθίε του. Επίση, δεν άκουσα να γίνεται λόγο για τον κοινωνικό αντίκτυπο στην, ε, ε, στην παρουσίασή σα. Øh, Ευχαριστώ για την παρουσίασή σα ενδιαφέρουσα η μελέτη. Να συμφωνήσω με αυτό που είπε ο Διευθυντής του ιδρύματο του Λιμπιλμπάου για τα θέματα της προστασία. Και να πω ότι ω ομάδα έχουμε υπάρξει ενθουσιώδης ω προ την παρουσίαση αυτή τη μελέτη. Και τις οδηγίες που αφορούν το πώς θα προσεγγίζουμε την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Νομίζω ότι πρέπει εδώ να πω ότι το θέμα είναι πώς θα μειώσουμε τον αριθμό των βιομηχανικών αντιστοιχημάτων κατά 25%. Αν έχουμε κατά 25% λιγότερους διοικητικούς κανόνες ως προς το διοικητικό φόρτο. Δεν νομίζω ότι αυτά τα δύο στοιχεία συνδυάζονται. Πιστεύω ότι στις εταιρείες όπου υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για, την, για τον εργαζομένο, εκεί υπάρχουν και καλύτερε επιδόσει. Νομίζω ότι οι χώρε επίση που επικεντρώνονται καλύτερα στο θέμα αυτό και το προστατεύουν καλύτερα έχουν και καλύτερα αποτελέσματα. Το λέω αυτό γιατί φαίνεται κάποια από τα πράγματα αυτά και εσείς ίδιοι να τα λάβατε υπόψη. Τώρα, ε, ανυπομονώ να μελετήσουμε με κάθε λεπτομέρεια αυτή την έκθεση, αλλά έχω κάποιες επιφυλάξεις Γιατί για τους ε, εργαζομένους με υψηλές δεξιότητες, με πολύ υψηλά προσόντα, πρέπει να σκεφτούμε πώς θα τους συγκρίνουμε με εκείνους που αντιμετωπίζουν πολλούς και σοβαρούς κινδύνους. Αυτό είναι κάτι που... Αυτό είναι ακριβώς που κοστίζει περισσότερο στην ε, κοινωνία μας. Μιλάμε για δισεκατομμύρια κορώνες, όταν υπάρχει ασθένεια που οφείλεται στι εργασιακέ συνθήκες ή κάποια μας στη δουλειά. Είναι και τραγικές πολλές φορές οι καταστάσει που προκύπτουν. Γι' αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σκεφτούμε τα πράγματα αυτά. Όταν θα φτάσουμε στην εξέταση τη οδηγία, δεν θέλουμε λιγότερου κανόνε για την υγεία και την ασφαλεία των εργαζομένων. Βεβαίω μπορούμε να έχουμε καλύτερου και βελτιωμένου κανόνε. Αλλά αν είχαμε περισσότερου κανόνε ίσω θα είχαμε καλύτερη υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Πριν σα δώσω πάλι το λόγο, ένα-δυο σχόλια και από μένα την ίδια. Προφανώ ικανοποιήθηκα ιδιαίτερω όταν είδα ότι μιλάτε για την υλοποίηση των οδηγιών. Αλλά θα ήθελα λίγα περισσότερα για τι συγκεκριμένε λεπτομέρειε, δηλαδή πώς ε, η οδηγία για τους εργαζομένους σε κατασκευαστικές εταιρείες, οικοδομές ε, θα υλοποιηθεί. Δηλαδή να δούμε την πραγματική υλοποίηση, στην πράξη, σε εταιρείε συγκεκριμένε. Έπειτα ήθελα να δω, ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν το έχει κάνει αυτό, μια επισκόπηση της υλοποίηση από το 2004. Ε, ξέρω ότι κάτι θα το έχουμε το 2013 στα χέρια μας, όμως πάντοτε θεωρώ ότι είναι πιο χρήσιμο να έχει κανείς συγκεκριμένα λεπτομεριακά στοιχεία παρά να κοιτάζει γενικώ ε, μάλλον τι γίνεται με συγκεκριμένους ε, με τους φυσικούς παράγοντες και τη σχετική οδηγία, με τη μείωση της επιχορύπανσης και πώς επηρέασε τις εταιρείες, ποια είναι το φέλη για τους εργαζομένους, η οδηγία για τις δονήσεις, παρομοίως, όλα αυτά τα καθοριστικά ζητήματα. Κάποια από αυτά είναι ιδιαίτερα περίπλοκα και αφορούν αμέσα του εργαζομένου. Αφορούν σίγουρα ένα μεγάλο φασματωμένο όμω τη δική μου τη σκοπιά. Θέλω να σα ρωτήσω αν πιστεύετε ότι η εντολή που σα δόθηκε, αυτό που σα ανατέθηκε να κάνετε, ήταν αρκετά συγκεκριμένο, αρκετά λεπτομερέ. Μήπω είχατε την αίσθηση ότι δεν μπορούσατε να τα εξετάσετε αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα, τι λεπτομέρειε τη υλοποίηση των πραγματικών οδηγιών στα πλαίσια αυτή τη μελέτη. Ήτανε κάποια απόφαση που τη λάβατε ίδια, η επιλογή. Έπειτα, για την αξιολόγηση κινδύνου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, δίνεται την εντύπωση, και αυτό κάπως μας προκάλεσε σύγχυση σε ορισμένα σημεία της μελέτης, σε κάποια σημεία φαίνεται να λέτε ότι η αξιολόγηση κινδύνου δεν είναι θέμα για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Ενώ σε κάποια άλλα σημεία λέει το αντίθετο. Επίση, αν δει κανεί τι μικρομεσαίες επιχειρήσει και πάλι και το τι πληροφόρηση έχουμε, έχουν για, την, ε, για το πώ πρέπει να υλοποιήσουν τι οδηγίε. Είναι καλή πληροφόρησή του. Αυτό πρέπει να εξετάσουμε, γιατί υπάρχουν εταιρείε που έχουν προβλήματα, ιδίω οι μικρέ, με αυτό ακριβώ το σημείο. Δεν μπορούν, δεν έχουν στα χέρια του όλο το διαθέσιμο υλικό. Δεν ξέρουν συγκεκριμένα τι να κάνουν με την καθοδηγία, τι λεπτομέρειε τη οδηγία. Χρειάζονται περισσότερη καθοδήγηση για να καταλάβουν ακριβώ τι πρέπει να προσέξουν και τι είναι το ζουμί, η ουσία. Ε, οι πληροφορίε λοιπόν για αυτό το θέμα ε, είναι, είναι αρκετά χρήσιμε. Ξέρω ότι προσπαθήσατε να συμπεριλάβετε κάτι για την καθοδήγηση για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Και ξέρω ότι δεν μα έχει μένει και πολλή χρόνο. Έχετε πάρα πολλέ ερωτήσει να απαντήσετε. Έχουμε και άλλη παρουσίαση μετά. Οπότε θα σα δώσω πέντε λεπτά. Πραγματικά σα παρακαλώ να παραμένετε στο πεντάλεπτο. Κάντε ό,τι μπορείτε να απαντήσετε στι ερωτήσει. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Ευχαριστώ. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να είμαι σύντομη. Πρώτα απ' όλα, δεν κατάλαβα το όνομα του πρώτου ομιλητού. Είπε ότι πρώτα πρέπει να ασχοληθούμε με την υγεία ασφάλεια των εργαζομένων και μετά με τα οικονομικά ωφέλη των εταιριών και επιχειρήσεων. Νομίζω αυτό είναι προφανέ. Όμω, η στόχευση τη μελέτη μα ήταν να δούμε αν μπορούμε να δείξουμε στι εταιρείε ότι υπάρχουν οικονομικά ωφέλη από το να ασχολούνται με το θέμα αυτό και να του δώσουμε περισσότερα κίνητρα, ώστε να επενδύσουν στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Αυτό ήταν ε, η σκοπιά μα, η προοπτική που ακολουθήσαμε στην έκθεση. Για του επιθεωρητέ, την επιθεώρηση και αν μπορεί να είναι πιο η όλη η διαδικασία, σίγουρα. Δώσαμε ένα παράδειγμα στην έκθεση. Για το σύστημα smile με χαμόγελα που χρησιμοποιείται στη Δανία. Εκεί χρησιμοποιούν ε, αυτές τις χαρούμενες, ή στενοχωρημένες φατσούλες ή αυτές που δεν έχουν ε, συγκεκριμένη έκφραση. Αυτό βοηθά να γίνει κάτι και βοηθά και τους επιθεωρητές της εργασίας ώστε να περάσουν σε διάλογο. Είναι επικοδομητικό αυτό. Δεν πρέπει κανεί να επικεντρώνεται στι κυρώσει, αλλά και στο πώ θα παρέχει συμβουλέ στι εταιρείε. Κάποιε από τι ερωτήσει φοβάμαι ότι δεν μπορώ να τι απαντήσω. Δεν έχω τι πληροφορίε. για την τηλεεργασία, την εργασία εξ αποστάσεω. Δεν ξέρω αν μπορώ να τα απαντήσω αυτά. Τώρα, για τα ψυχοπαθολογικά προβλήματα και το επίπεδο κοινωνικού διαλόγου στην εταιρεία, τον συσχετισμό που ζητήσατε. Σίγουρα υπάρχει συσχετισμό. Όμω δεν έχω τι πληροφορίε για να απαντήσω. Δεν μπορώ να απαντήσω ούτε σε αυτό. Για τον κύριο Κρίστενσεν. Μα ρωτήσατε εάν μπορεί κανεί να τεκμηριώσει ότι οι εταιρείε που επενδύουν στα ζητήματα που μα απασχολούν έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό ξεκινήσαμε να κάνουμε, αλλά όπω είπα, ε, υπάρχει ανάγκη για περισσότερη έρευνα σε αυτόν τον τομέα. Κάποια τεκμηρίωση υπάρχει. Βλέπουμε ότι αν κανείς επενδύει στην εργασιακή ασφάλεια και υγεία υπάρχει μια αύξηση των επιδόσεων, όμως δεν ε, είναι αρκετά τα στοιχεία ούτε πολυπιστικά για τη διεύθυνση των επιχειρήσεων. Έπειτα. Κυρία Λίν, πολύ γρήγορα τις είπατε τις ερωτήσεις σας. Είπατε ότι θα θέλατε να έχουμε προχωρήσει περισσότερο προς την υλοποίηση στην πράξη των οδηγιών, όλων των οδηγιών. Και ε, ρωτήσατε αν η εντολή, αυτό, η, ευθύνη, η έρευνα που ανατέθηκε ήταν πολύ συγκεκριμένη ή όχι. Να πω ότι θα έπρεπε να έχουμε επιλέξει συγκεκριμένε οδηγίε για να περάσουμε σε πάρα πολλέ λεπτομέρειε. Αλλά ακόμα και έτσι θα χρειαζόταν μια ακόμη μεγαλύτερη μελέτη και πολύ περισσότερη πόρη για να εκπονηθεί. Νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν ενδιαφέρον να γίνει αυτό, αλλά δεν ήταν εφικτό εντό τη εντολή για τη μελέτη αυτή. Επίση, είπατε ότι δεν είναι σαφέ εάν η εξολόγηση του κινδύνου είναι ένα πρόβλημα για τι μικρομεσαίε ή όχι. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ναι, είναι πρόβλημα για κάποιε μικρομεσαίε. Αλλά και για άλλου φαντάζομαι, θα συμφωνείτε έτσι. Δεν φαντάζομαι να διαφορετική απάντηση. Έπειτα, οι πληροφορίε για την υλοποίηση των οδηγιών προ τι εταιρείε χρειάζονται περισσότερη καθοδήγηση. Ναι, νομίζω σαφώ χρειάζονται περισσότερη. Αναφέρθηκε ότι ένα, μια από τι προτάσει για τη μείωση του διοικητικού φόρτου ακριβώ ασχολείται με την παροχή καλύτερη καθοδήγηση στις κατασκευαστικές εταιρείες. Νομίζω είναι σαφές ότι χρειάζεται αυξημένη καθοδήγηση εδώ, ιδίως στους τομείς του κινδύνου. Νομίζω θα σταματήσω εδώ. Υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις, αλλά δεν μπορώ να τις απαντήσω τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να σας ευχαριστήσω που ήρθατε και κάνατε αυτή την παρουσίαση. Σα ευχαριστούμε ιδιαίτερως. Επόμενο σημείο, η ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Σταϊνμπούκα, διευθυντή της Eurostat για τους ε, δείκτες της ένδυας. Σας δίνω κατευθείαν το λόγο. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερος. Thank you very much, for... Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα να ζητήσω από τους τεχνικούς ε, να φορτώσουν την παρουσίασή μου. Είναι πολύ μεγάλη τιμή και χαρά για μένα να συμμετέχω στη σημερινή σας συνεδρίαση. Μπορώ και να ακούσω αυτά που λέτε, αλλά μπορώ επίσης ε, να συνεισφέρω σε σχέση με την συμβολή της Eurostat για την μέτρηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης ε, στην Ευρώπη. Μία παρατήρηση μόνο θα ήθελα να κάνω. Ήμουν διευθύντρια οικονομικών και περιφερειακών στατιστικών, αλλά τώρα είμαι διευθύντρια ε, στατιστικών που αφορούν ε, την ε, κοινωνία των πληροφοριών. Οπότε, απλώς το επισημαίνω για να το γνωρίσετε. Περιμένω την παρουσίασή μου να φορτωθεί πριν αρχίσω. Ναι, περιμένουμε οι τεχνικοί να εμφανίσουν την παρουσίαση. Yeah, okay, it's back again. Ωραία. Συνήθως αλλάζω μόνη μου τις διαφάνειες, αλλά όχι σήμερα. Οπότε με λιγάκι από τη δική σας ε, συνδρομή. Επόμενη διαφάνεια. Είναι πολύ μεγάλη πρόκληση για τις κοινωνικές στατιστικές στην Ευρώπη η μέτρηση του, της προσπάθειας που πρέπει να γίνει από την φτώχεια στην κοινωνική ενσωμάτωση. Γιατί εμείς πρέπει να παρέχουμε στους διαμορφωτές πολιτικής αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας στατιστικές που δίνουν σαφή εικόνα για το κατά πόσο οι ευρωπαϊκές χώρες κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή από τη φτώχεια στην κοινωνική ενσωμάτωση και όχι αντιστρόφως. Υπάρχουν ε, πάρα πολλοί μοχλοί ε, στη Eurostat. Καταρχάς θα ήθελα να αναφερθώ στην ε, στρατηγική της Ευρώπης για το 2020 που αναφέρει ειδικότερα στην φτώχεια και την κοινωνική ενσωμάτωση και δεν αναφέρεται βέβαια μόνο σε αυτά τα θέματα, αναφέρεται και στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας και όλα αυτά τα στοιχεία, αν όχι άμεσα, έμεσα συνδέονται με την κοινωνική ενσωμάτωση. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στο, στην ανακοίνωση ΑΕΠ και πέρα από αυτό που δίνει σαφή εντολή στην Eurostat και ένα σαφή προσανατολισμό σε σχέση με τη μέτρηση των κοινωνικών δικτών με ιδιαίτερη έμφαση στη μέτρηση των ανισοτήτων στις ευρωπαϊκές οικονομίες, κοινωνίες, συγγνώμη, όπως επίσης και στο ειδικό αίτημα αύξησης του έγκαιρου των στατιστικών. Θα ήθελα να αναφερθώ επίσης ε, στην Επιτροπή Stiglitz ε, και την ε, πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Σαρκοζή, γιατί οι συστάσεις αυτές που συμπεριλαμβάνονται μας δίνουν πολύ καλύτερες πληροφορίες για το πώς μπορούμε καλύτερα να προσμετρήσουμε τις ανισότητες. Και τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, η πίεση ε, λόγω της ε, συνεχιζόμενης κρίσης δίνει ακόμη μεγαλύτερη όθηση στους ε, στατιστικολόγους κοινωνικών στατιστικών για να μετρήσουν καλύτερα το πώς έχουν τα πράγματα σε σχέση με τη φτώχεια και την κοινωνική ενσωμάτωση, κάτι που επιδεινώθηκε ιδιαίτερως κατά τη διάρκεια της κρίσης. Επόμενη διαφάνεια. Στις κοινωνικές στατιστικές εμείς ε, παρέχουμε πολλούς δείκτες, ε, πολλούς τρόπους μέτρησης της κοινωνικής διάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δείκτες που ανέφερα κανονικά ε, καταγράφουν την πρόοδο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το 2020 ε, και ειδικότερα υπάρχουν θεματικές ενότητες επί των οποίων επικεντρωνόμαστε. Θα ήθελα όμως να αναφέρω και πολλούς άλλους δείκτες οι οποίοι είναι ήδη στη διάθεσή μας στο πλαίσιο της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού για την ε, ε, κοινωνική ενσωμάτωση και την κοινωνική προστασία. Οι δείκτες αυτοί ορίζονται από την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας και μπορούν να προτείνουν και άλλους δείκτες πολύ πιο περιεκτικούς για την κοινωνική διάσταση, για τις τάσεις των συντάξεων, ε, για την υγεία για την ε, φροντίδα, την ιατροφαρμακευτική περίθελψη. Υπάρχουν λοιπόν δείκτες σε πάρα πολλά επίπεδα, δεν μπορώ να τους αναφέρω όλους, πάντως υπάρχουν και χρησιμοποιούνται ε, ενεργά στο πλαίσιο της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού. Επόμενη διαφάνεια. Έχουμε ακόμη ορισμένα εκρεμή ζητήματα και προκλήσεις ε, ενώπιών μας, γιατί θέλουμε να μετρούμε καλύτερα την, ε, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την φτώχεια. Και για να το επιτύχουμε αυτό πρέπει να είμαστε σαφείς ως προς τον ορισμό του κοινωνικού αποκλεισμού. Και θα ήθελα να αναφερθώ στο 1995, στον ορισμό του Συμβουλίου το 1995 για τον κοινωνικό αποκλεισμό, άτομα, οικογένειες και ομάδες των οποίων οι πόροι ε, ηλική και κοινωνική είναι τόσο περιορισμένοι ούτως ώστε να τους αποκλείουν από τον αποδεκτό τρόπο διαβίωσης το κράτος μέλος το οποίο διαμένουν. Αυτός είναι ένας γενικός ορισμός. Όμως το ζήτημα είναι πώς μπορούμε να το μετρήσουμε αυτό, πώς μπορούμε αυτήν την ποιοτική, τον ποιοτικό ορισμό να τον μεταφράσουμε σε κάτι ποσοτικό. Η πρόκληση λοιπόν που προκύπτει για μας είναι να μετρήσουμε τις διάφορες διαστάσεις ε, του κοινωνικού αποκλεισμού με ένα σύνολο δικτών. Είναι αδύνατον να έχουμε έναν δείκτη ή δύο δείκτες ή ένα, ένα σύνολο και μόνο δικτών που μας βοηθούν να μετρήσουμε όλες τις διατάσεις του, κοινωνικού αποκλεισμού. Για παράδειγμα η κατάσταση της αγοράς εργασίας, η φτώχεια, η κοινωνική προστασία, η υγεία, η εκπαίδευση, πρόσβαση σε δημόσιες ιδιωτικές υπηρεσίες, στέγαση, ε, δικαιώματα του πολίτη, κινητικότητα, ε, κοινωνική και πολιτική συμμετοχή, αναψυχή, ε, πολιτιστικές δραστηριότητες. Δεν είναι διεξοδικός ο κατάλογος όλων αυτών των διαστάσεων που σας ανέφερα, βάσει των οποίων μπορούμε να μετρήσουμε σωστά ε, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Όπως καταλαβαίνετε, χρειαζόμαστε ένα σύνολο δικτών πρέπει να μπορούμε να προσμετρήσουμε την κατάσταση όπως εξελίσσεται. Χρειαζόμαστε δηλαδή τάσεις και χρειαζόμαστε όλες αυτούς, όλους αυτούς λοιπόν τους δείκτες ε, με κατανομή ανακατηγορία. Και θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή ότι οι κατηγορίες και οι διαστάσεις είναι διαφορετικό πράγμα. Όταν μιλάω για κατηγορίες, μιλάω για το φύλλο, την ηλικία, διάφορες κατηγορίες λοιπόν πληθυσμού. Ένα πολύ σημαντικό σημείο που για να μετρήσουμε την ένδυα μέσα στο χρόνο είναι ότι σε όλες τις ε, κοινωνίες και στις ευρωπαϊκές χώρες επίσης υπάρχουν κατηγορίες μάλλον μόνιμες ή έμονες λέει ο Μιλήτρια ε, ανθρώπων ως προς την γραμμή της φτώχειας και δεν ξέρουμε αν αυτή η αιμονή θα διατηρηθεί ή αν θα μπορέσουν να μειωθούν αυτές οι κατηγορίες στο στον ελάχιστο μόνο δυνατό βαθμό. Κάθε δείκτης εδώ θα πρέπει να είναι δείκτης υψηλής ποιότητας, διότι κάθε πληροφορία προσφέρουμε στους ε, αρμόδιους για των αποφάσεων, για τη χάραξη πολιτικής πρέπει να είναι σαφής, έγκαιρες, ακριβής, διαρκής και εύστοχες. Εάν λοιπόν δεν το καταφέρουμε αυτό, θα έλεγα πρόκειται για μολυσμένες πληροφορίες, τότε δεν έχουμε καταφέρει τίποτα. Και κάτι ακόμη. Έχουμε αναπτύξει ε, τις ενοιολογικές μας διαστάσεις ε, ως προς τον κίνδυνο της φτώχειας, την ε, στέρηση υλικών αγαθών και το κακό επίπεδο στέγης. Αυτοί είναι οι τρεις ε, παράγοντες που έχουμε προσδιορίσει, τρεις κατηγορίες αν θέλετε και ε, συνεργαζόμαστε στενά και με την Eurostat προκειμένου να, προσδιορίσουμε, να αξιοποιήσουμε μάλλον αυτούς τους δείκτες. Εδώ έχουμε μέτρηση σε ατομικό επίπεδο, επίπεδο νοικοκυριού προκειμένου να καταγραφούν και οι ανισότητες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι δηλαδή μέση δείκτη, δείκτες, δείκτες μέσης χρήσης. Δεν μπορούμε να πούμε ότι Φερρυπίν καταγράφουμε μία μέση θερμοκρασία για τα νοσοκομεία. Όχι, έχουμε δείκτες ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Και επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η διαφορετική... Ε, διαφορετικές συνιστώσεις είναι καλύτερη από τους διαφορετικούς ε, δείκτες, γιατί όταν γίνεται επιλογή δικτών ε, υπησέρχονται υποκειμενικές κρίσεις. Δεν μπορεί να είναι απόλυτα ε, αμερόληπτη η κρίση της φτώχειας, γι' αυτό προτιμούμε να έχουμε τρεις διαφορετικούς δείκτες, λέει η ομιλητρία. Θα ήθελα τώρα να σας περιγράψω έναν προς έναν αυτούς τους δείκτες. Καταρχάς έχουμε τον κίνδυνο της φτώχειας. Εδώ δηλαδή έχουμε να κάνουμε με επίπεδο χαμηλότερο από το 6% του μέσου όρου, θα σας το δείξω, και μετά έχουμε και μια κατανομή ένα χώρα στην επόμενη ε, διαφάνεια βλέπετε ε, τι ακριβώς εννοούμε, δηλαδή μπορείτε να δείτε την κατανομή εισοδήματος με λογαριθμική κλίμακα, λογαριθμική κλίμακα γιατί, διότι διαφορετικά η ορατότητα με τις στήλες θα ήταν πολύ ε, επιβαρημένη, θα ήταν πολύ κακή. παίρνουμε λοιπόν μετά την το μέσο όρο αυτής της κατανομής εισοδήματος και προχωρώντας στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε ότι έχουμε 60% αυτού του μέσου όρου που καταγράφει το 60% του εισοδήματος αυτού του πληθυσμού στην Ευρώπη. Και συνεχίζουμε για να πούμε ότι μας ενδιαφέρει στα αριστερά σας, στα αριστερά της διαφάνειας μάλλον το τμήμα που δείχνει ανθρώπους οι οποίοι ζουν κάτω από το ποσοστό φτώχειας, που είναι η πραγματικά φτωχή. Και έτσι καταγράφοντας αυτούς τους ανθρώπους, υπολογίζουμε ότι είναι το 20% του ευρωπαϊκού πληθυσμού και 20% σε κίνδυνο φτώχειας. Και επίσης βλέπετε τις τάσεις του τμήματος του πληθυσμού. δεν έχουμε να κάνουμε δηλαδή με το πιο ευάλωτο πληθυσμό στην Ευρώπη. Συνεχίζουμε με τον ίδιο πάλι αλλά με κατανομή στις χώρες, αναχώρα. Βλέπετε το ποσοστό φτώχειας από το αριστερό τμήμα της διαφάνειας με την τσεχική δημοκρατία μέχρι το δεξί τμήμα που είναι η Λετωνία. Δεν ξέρω αν μπορείτε να τα αρχικά των κρατών αλλά πάντως εμείς θελήσαμε να καταγράψουμε τον, το ποσοστό του κινδύνου φτώχειας σε σύγκριση με το κατόφλι του κινδύνου φτώχειας. Γιατί εδώ έχουμε διαφορά. Και βλέπετε ότι για την κάθε χώρα το κατόφλι είναι διαφορετικό. Σε ορισμένες χώρες είναι πολύ χαμηλό το κατόφλι, όπως η Ρουμανία, Φερρυπίν, που είναι η δεύτερη από τα αριστερά, με κατόφλι χαμηλό μένα, αλλά και κίνδυνο, ποσοστό δηλαδή κινδύνου να περιπέσει κανείς σε συνθήκες φτώχειας, πάρα πολύ ψηλό, πολύ ψηλότερο δηλαδή από το κατόφλι. Ενώ για την Τσεχική Δημοκρατία που είναι η πρώτη χώρα από τα αριστερά μας, ο κίνδυνος της φτώχειας είναι πολύ χαμηλότερος από τη, για τη Ρουμανία παραδείγματι, γιατί είναι χαμηλότερος από το κατόφλι. Το κατόφλι όμως πράγματι εξαρτάται από τα όρια που έχει η κάθε χώρα και ελπίζω να έχουν επιλεγεί ε, σωστά ε, και στις διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνεχίζω. Κίνδυνος φτώχειας αναφύλλω. Δίνουμε δηλαδή, όπως είπα, πληροφορίες ανακατηγορία πληθυσμού. Και θα δείτε πάλι άνδρες και γυναίκες με κίνδυνο φτώχειας στις ευρωπαϊκές χώρες. Ελπίζω να σε αφήσει οι διαφάνειές μου και πάνω απ' όλα ελπίζω να μπορέσω να τις έχω σε αντίγραφα έτσι ώστε να τα δείτε και εσείς. Έχουμε φέρει βέβαια κάποιες, ε, κάποια φυλάδια στην είσοδο της ε, αίθουσας για τη φτώχεια αλλά δεν είναι τόσο πολλά ίσως. Συνεχίζω με τον κίνδυνο φτώχειας σε κατανομή ηλικίας, ομάδας ηλικίας, όπου θα ήθελα να υπογραμμίσω τον κίνδυνο της φτώχειας για τα παιδιά, ηλικίας κατά το 18 και τους ηλικιωμένους. Ηλικία ανά των 60. Βλέπετε λοιπόν αυτούς τους κινδύνους, αυτές τις ε, ομάδες τις πιο ευάλωτες και τον κίνδυνο της ε, φτώχειας. Ε, συνεχίζω με τον κίνδυνο φτώχειας και την αιμονή ή την μονιμότητα του κινδύνου που πάλι διαφέρει αναχώρα. χώρα. Εδώ δεν έχουμε τα στοιχεία για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά για τις περισσότερες εξ αυτών. Και φαντάζομαι θα βρείτε στη διαφάνεια ότι υπάρχει μια επιλογή κρατών ε, αρκετά αντιπροσωπευτική. Προχωρώ τώρα με τον επόμενο δείκτη για την προσμέτρηση της φτώχειας και της, το κοινωνικό αποστέρηση από υλικά αγαθά άτομα δηλαδή ή νοικοκυριά τα οποία από ένα κάνιστρο εννέα αγαθών δεν διαθέτουν τα τρία. Φερρυπίν, διακοπές, αυτοκίνητο, ε, τουαλέτα και κατάλληλο εξοπλισμό ε, υγιεινής, ε, στέγη, σωστή δηλαδή μπορεί να μπάζει νερά, η στέγη, η τύχη κτλ. Και αυτά και άλλα τέτοια, ε, όπου όμως πάλι είναι διαφορετική η κατάσταση ανά χώρα, γιατί είναι διαφορετική η εικόνα που προσφέρει η Ρουμανία σχέση με το Λουξεμβούργο, Φερρυπίνη, το Βέλγιο, με αυτό τον δείκτη. Και πάλι για, την, ε, ε, για τους δείκτες της Ευρώπης 2020 έχουμε ορίσει ότι η σοβαρή αποστέρηση από υλικά αγαθά θα οριστεί στα 4 εκ των 9 που έχουμε προσδιορίσει στο κανέστρο και εφόσον λείπουν αυτά θα ε, συμπεραίνουμε ότι προσπρόκειται για βαρία αποστέρηση από αγαθά. Και μετά βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζουμε αυτή την ε, μονάδα, την αποστέρηση δηλαδή ε, υλικών αγαθών μεγάλες αποκλήσεις έχουμε από το Λουξεμβούργο μέχρι τη Βουλγαρία. Θα φαντάζεστε και εσείς ότι το Λουξεμβούργο είναι στα αριστερά, στα δεξιά μα της διαφάνειας βρίσκεται η Βουλγαρία. Και η στήλη που βλέπετε στα, στην άκρη αριστερά της ε, διαφάνειας είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεχίζω με έναν άλλο δείκτη που είναι η χαμηλή ένταση εργασίας, δηλαδή ότι απασχολείται κανείς σε ποσοστό κάτω του 20% των εργασιακών του δυνατοτήτων. Μπορούμε να προσμετρήσουμε λοιπόν αυτό το ποσοστό και έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που ζουν σε νοικοκυρία χαμηλής έντασης εργασίας και πάλι βλέπουμε από την αριστερά, στην αριστερή πλευρά την Κύπρο, στη δεξιά την Ιρλανδία. Ίσως δεν είναι εύκολο να συγκριθούν αυτοί οι δείκτες. Αλλά αν προχωρήσουμε στην επόμενη διαφάνεια, θα έλεγα ότι τη φτώχεια δεν μπορούμε να την προσμετρήσουμε στην Ευρώπη με ένα μόνο δείκτη, γιατί και οι τρεις δείκτες δίνουν μάλλον αντιφατικές μεταξύ τους εικόνες. Επικράτονται σε ένα βαθμό, αλλά όχι 100% δεν ταυτίζονται. Και γι' αυτό προσπαθούμε να βρούμε τα κοινά σημεία, αυτή για να δούμε την εικόνα της Ευρώπης των 27. Με το ροζ είναι ο κίνδυνος της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού. Όχι, διορθώνει ο Μιλήτρια. Ο κίνδυνος της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού εκφράζει το συνολικό αριθμό που μπορούμε να υπολογίζουμε αποκλείοντας από τους υπολογισμούς μας τα επικαλυπτόμενα σημεία. 115 εκατομμύρια πολίτες της Ευρώπης. Αφορά αυτό το θέμα. Στο ροζ, λοιπόν, έχουμε τον κίνδυνο της φτώχειας, δηλαδή 81 εκατομμύρια. Στο πράσινο έχουμε την ε, βαρία αποστέρηση με 41 εκατομμύρια. Και στο, μπλε τα νοικοκυριά τι εργασίε με 31 εκατομμύρια πολίτε. Έτσι, αν θέλουμε, όπω βλέπετε, μηχανικά, καθαρά, μηχανιστικά καθαρά να καταμετρήσουμε αυτόν τον πληθυσμό, μπορούμε ε, να το πράξουμε εφόσον αποκλείσουμε τα σημεία επικάλυψης. Αν όμω δεν χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μέθοδο, τότε μόνο εν μέρη θα έχουμε καταγράψει τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να συνδυαστούν τα τρία αυτά ε, οι τρεις αυτοί τρόποι μέτρησης. Και συνεχίζω στην επόμενη διαφάνεια, που είναι μάλλον αντίστοιχη. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω τον συνδυασμό των δικτών αυτών και να πω ότι διαφέρει πολύ πάλι αναχώρα. Κοιτώντας τα αριστερά της διαφάνειας. Προκτήρια για την ίδια διαφάνεια που είδαμε μόλις τώρα. Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσος όρος. Στα δεξιά και πάνω έχουμε τις κάτω χώρες. Στις κάτω χώρες λοιπόν η αποστέρηση από υλικά αγαθά είναι μάλλον περιθωριακή. Ο κίνδυνος όμως φτώχειας και η χαμηλή ένταση εργασίας είναι μάλλον υψηλή και έτσι ο συνδυασμός του ροζ και του μπλε μαζί μας δίνει το μεγαλύτερο τμήμα των, πολιτών, των ανθρώπων εκείνων που αντιμετωπίζουν αυτό το φαινόμενο. Μια διαφορετική εικόνα μας δίνει η Ρουμανία τώρα που βλέπετε ότι το ροζ χρώμα και το πράσινο με την ε, βαρύ αποστερήση από αγαθά και είναι πολύ μεγάλο κομμάτι, όπως και ο κοινωνικός αποκλεισμός, ενώ το μπλε κομμάτι που είναι η χαμηλή ένταση εργασίας στο νοικοκυριό είναι μάλλον μικρό ως δείκτης. Και πάλι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να συνδυάσουμε τους τρεις αυτούς δείκτες. για να μπορέσουμε να καταμετρήσουμε Πλήρω του φτωχού. Και κλείνω τώρα με, την, με τα συμπεράσματα στη τελευταία μου διαφάνεια. Ο κοινωνικό αποκλεισμό και φτώχεια επηρεάζει πολλά τμήματα και υπό του πληθυσμού. Δεν υπάρχει ένας δείκτης, ε, για να, ένας για να προσμετρηθεί. Έτσι λοιπόν ένα ισορροπημένο και καλά οργανωμένο χαρτοφυλάκιο δικτών απαιτείται να εξευρεθεί έτσι ώστε αυτοί που κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό να καταγραφούν με βάση τους τρεις δείκτες της φτώχειας και, του, και της φτώχειας, της και της αποστέρησης από υλικά αγαθά. Βεβαίω αυτά χρησιμοποιούμε και ταυτόχρονα προσπαθούμε να βελτιώσουμε τι συνθήκε τις τις συνθήκες καταγραφή, συγγνώμη, την έγκαιρη συλλογή των στοιχείων, όπου πάλι έχουμε βέβαια δυσκολίε και η επόμενη ε, κατάθεση προτάσεων, ε, στοιχείων μάλλον, να προβλέπεται για φέτος, ακόμα τον Νοέμβριο, δηλαδή μέσα στο μήνα. Η προηγούμενη πρόταση ήταν του 2009. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Είμαστε θέση σας για οποιαδήποτε ερώτηση υπάρχει και για να ακούσω φυσικά τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ. Thank you very much. I found that very Ευχαριστούμε πολύ. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα παρουσίαση άκρος χρήσιμη. Κυρία Σουέτερ. Ευχαριστώ. Η πρότασή μου έχει να κάνει με το γεγονό ότι Έχοντα μιλήσει με την Επιτροπή στην Κλίτση, είχαμε πει ότι χρειάζονται αυτοί οι δείκτε για να υπολογιστεί η πρόοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, το 2020. Αλλά αυτό το αμφισβητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι χρειάζονται οι δείκτε αυτοί. Και γι' αυτό, γιατί λέτε ότι δεν μπορούν να καταγραφούν ακόμα, δεν υπάρχουν οι μέθοδοι. Δεν υπάρχουν αρκετά συγκρίσιμες μέθοδοι για να συλλέξουμε τα στοιχεία αυτά. Και γι' αυτό ρωτώ εάν τα στοιχεία τα οποία μας δώσανε τώρα με βάση τους τρεις δείκτες επιτρέπουν την ε, χρήση μεθόδων ε, τυποποιημένων, εάν μπορούμε δηλαδή να τα αξιοποιήσουμε πράγματι, αν έχετε εντοπίσει τη χρησιμότητά τους, ή αν υπάρχει κάτι άλλο κατά την άποψη σας που χρειάζεται για να αξιολογήσουμε την κοινωνική ενσωμάτωση, για να εξασφαλίσουμε την, ε, για να προσμετρήσουμε την διαχείριση της φτώχειας. Ευχαριστώ κυρία Τσίμερ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση των δικτών εν γέννη και ιδιαίτερα των συμπερασμάτων στα οποία θα πρέπει να καταλήξουμε και του προσδιορισμού της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020 και τον καλύτερο προσδορισμό, τον υπολογισμό μάλλον της φτώχειας. Η φτώχεια από ό,τι βλέπω στα κράτη είναι διαφορετική, αυτό το ξέραμε τους ή άλλους αλλά ταυτόχρονα έχουμε να κάνουμε και με τη φτώχεια, η οποία μέσα σε ένα κράτο στην περιφέρεια ενό κράτου έχει διαφορετική παρουσία, διαφορετική εικόνα και πρέπει να, με, να καταμετρηθεί μάλλον με διαφορετικό τρόπο και ανάλογα με το ει κατηγορίε του πληθυσμού ή ανάλογα με τι περιφέρειε. Όλα αυτά μου φαίνονται πολύ λογικά και σαφή. Αυτό που δεν είναι τόσο σαφέ για μένα και δεν μπόρεσα να καταλάβω τόσο καλά με την παρουσίασή σα. Είναι το εξής μας εξηγήσατε ότι είναι σημαντική η διασύνδεση των τριών δικτών για να μπορέσουμε να καταγράψουμε τη φτώχεια κατά τρόπο διαφοροποιημένο και αντίστοιχα να προτείνουμε μέτρα. Όμως, Όταν μας λένε οι Υπουργοί των Κοινωνικών Υποθέσεων των κρατών μελών ότι κάθε κράτος έχει τη δική του Ε, συλλογή δικτών ή πρέπει μόνο του να προσδιορίσει τους δείκτες του. Πώς να το καταλάβω εγώ αυτό. Δηλαδή η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας ε, άκουσε πριν από ε, λίγες μέρες από τον Υπουργό του να λέει ενώπιον του Κοινοβουλίου ότι θα έχει δείκτη ο οποίος θα υπολογίζει, θα προσμετρά την μακροπρόθεσμη ανεργία σε έναν οικοκυριό. Αυτός ο δείκτης πώς θα συνδυαστεί ή πώς πρέπει να συνδυαστεί κατά την με τους άλλους γιατί μην ξεχνάμε ότι με τη στρατηγική 2020 έχουμε δεσμευθεί να μειώσουμε κατά 20% τη φτώχεια εκείνων οι οποίοι έχουν μείνει μακροχρόνια άνεργοι, βρίσκονται σε νοικοκυριό με μακροχρόνια φαινόμενο ανεργία. Αυτή είναι η ερώτηση στην οποία δεν έλαβα απάντηση ε, από την παρουσία σας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μωρέ Σαρτιέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η πρώτη μου ερώτηση αφορά Αυτά ε, που είπε η κυρία Τσίμερ για, την, ε, για τους δείκτες αναχώρα και θα ήθελα να προσθέσω το εξής. Μήπως θα μπορούσαν οι, χώροι, οι χώρες να διαλέξουν ε, διαφορετικούς δείκτες, αλλά ακόμη παραπέρα, ακόμη πέρα από αυτό, μήπως μπορούμε καλύτερα να διαλέξουμε τους δείκτες, τους ορισμούς των δικτών από τη μία χώρα στην άλλη. Το περιεχόμενο των δικτών είναι ίδιο από τη μία χώρα στην άλλη. Γιατί αν θέλουμε να μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις μεταξύ ε, κρατών, πρέπει να συμφωνούμε επί του περιεχομένου του δείκτη. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη μου ερώτηση είναι η εξής. Βλέπουμε πόσο ενδιαφέροντα γίνονται, γίνονται όλα όταν χρησιμοποιείτε τις στατιστικές σας ε, για ομάδες τύπου άνδρες-γυναίκες ή δημογραφικές ομάδες, δηλαδή ανάλογα με την ηλικία, προκειμένου οι δείκτες και τα αποτελέσματα από τους δείκτες ε, γιατί από τους δείκτες μόνους τους δεν μπορούμε να βγάλουμε κανένα συμπέρασμα. Για να μπορέσουμε λοιπόν να αναλύσουμε τους δείκτες αυτούς ε, και να λάβουμε αποφάσεις τι μας λείπει. Τι μας λείπει σήμερα για να μπορούμε να έχουμε κάποια στοιχεία που θα μπορέσουν να επηρεάσουν τις πολιτικές και τις αποφάσεις μας στο μέλλον. Δηλαδή, ο συνδυασμός των δικτών επαρκεί. Και η τρίτη μου ερώτηση είναι η εξής. τη μετακίνηση της φτώχειας, τη γεωγραφική πώς την μετράτε. Δηλαδή βλέπουμε χώρες ε, της Ευρώπης ε, στις οποίες η φτώχεια η σημαντική, το σημαντικό επίπεδο στο, ε, φτώχειας είναι περίπου ο μέσος όρος. Βλέπουμε μετακίνηση του πληθυσμού από την Ήπεθρο στο Άστι. Κατά τη γνώμη σας, πώς μπορεί ακριβώς να προσμετρηθεί το φαινόμενο αυτό κυρία Τόνα. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Δύο ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, το θέμα της ένδυας, όπως προσέστε στην, στο φυλάδι αυτό. Ποια είναι η μέθοδό σας για τα θέματα αυτά, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον και από αυτήν την άποψη το συγκεκριμένο ζήτημα. Επίση για τι εξελάξεις, εγώ προηγουμένω δεν έχω, για τις εξελίξεις δεν έχω ξαναδεί τέτοιε στατιστικέ. Μιλάμε για αριθμού το 2009. Έχετε αριθμού και για, άλλους, για άλλες χρονιές. Και έπειτα εδώ υπάρχει ένα δίλημα. Υπάρχει κρίση απασχόληση στην Ευρώπη, πολλοί είναι άνεργοι, οπότε αν επιστρέψουν στην εργασία, εάν αυξηθεί η επιστροφή στην αγορά εργασία, μπορεί να αυξηθούν και ανισότητε. Μπορείτε να πείτε δύο λόγια και για αυτό το δίλημα. Διότι όταν κάποιοι περνάνε πια στην ε, ενεργοδράση, πάλι οι κοινωνικέ διαφορέ αυξάνονται. Έχετε λοιπόν κρατήσει τι αναλογίε στην καταμέτρηση τη ένδυα. Μπορείτε να το λάβετε αυτό υπόψη στις μετρήσεις σας, διότι κάποιοι, ε, φόσον επιστρέψουν στη δουλειά, κάποιοι άλλοι θα γίνουν ακόμα φτωχότεροι σε σχέση με αυτούς. Πώς το μετράμε αυτό. Ευχαριστώ. Πριν σας δώσω πάλι το λόγο, και εγώ έχω μια-δυο παρατηρήσεις. Όπω και άλλοι για, που παρα, έκαναν παρατηρήσει για διάφορου δείκτε και διάφορα θέλω και εγώ να πω. Ε, πιστεύετε ότι θα υπάρξει πρόβλημα όταν το εξετάσατε, γιατί εγώ θα τον πίνακά σα και εσεί αναφέρετε τρία από τα στοιχεία που νομίζω ότι συνολικά ήταν εννιά για τον ορισμό τη φτώχεια. Μιλάμε για το αυτοκίνητο, για το πλυντήριο. Εγώ αυτό δεν νομίζω ότι είναι το ίδιο με μια στέγη που στάζει και άλλα πολλά από τον κατάλογο. Δεν έχουμε μάλλον διερμηνία σε μια από τις γλώσσες, τα γαλλικά κατά πάσα πιθανότητα. Να συνεχίσω, εντάξει. Μας ακούτε? Έχετε διερμηνία, κύριε Γκρινέ. Μάλιστα. Όπως έλεγα, το αυτοκίνητο και το πλυντήριο σε κάποια κράτη-μέλη δεν νομίζω ότι μπορεί να τα ορίσει κανείς την απουσία του ως φτώχεια. Ενώ σε περισσότερα κράτη-μέλη μπορεί να ίσχυε κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η δυσκολία. Όταν τα συμπεριλαμβάνεται στον ίδιο κατάλογο με τη στέχη που στάζει και όλα τα υπόλοιπα που αναφέρεται, Έπειτα. Επίση για άλλου τομεί τη απασχόληση από τα γραφικέ επαναστάσει, εδώ διάφορε χώρε έχουν πολύ συγκεκριμένε οργαν... Ε, οργανώσει για τους ε, για τα, μάλλον ότι μετράτε τα νοικοκυριά των εργαζομένων. Σε κάποια μέλη όμω οι συνθήκε για αυτά τα νοικοκυριά είναι τελείω διαφορετικέ. Δεν υπάρχει αυτή η έννοια. Οπότε βλέποντα τα πράγματα ανακάτω μέλο αλλάζει πολύ η εικόνα. Επειδή λοιπόν έχουν τέτοιε οργανώσει κάποια κράτη-μέλη, επιλέγουν του δείκτε, άρα το να μετατοπίσουμε του δείκτε από 100 μέλο σε 100 μέλο δεν δείχνει απαραίτητα την σχέση μεταξύ όλων. Για τη διάκριση τώρα, τη κριτική συμπεριφορά. Υπάρχει κάτι ε, σε σχέση με ένα δείκτη που να ορίζει πώ η διάκριση επηρεάζει τον κοινωνικό αποκλεισμό. Γνωρίζω από την σκοπιά των ε, ηλικιωμένων πολιτών Υπήρχε για εδώ και μια γραφική παράσταση. Οι ηλικιωμένοι ακριβώ άνθρωποι μαζί με τα παιδιά σε κάποια κατημέλη βάσει τη γραφική σα παράσταση τείνουν να βρίσκονται σε συνθήκε ένδυα. Υπάρχει όμω κανένα δείκτη του κοινωνικού αποκλειτισμού για του ηλικιωμένου και του ανθρώπου με ειδικέ ανάγκε. Είδα από την παρουσίασή σα ότι Υπάρχει διάσταση στο κοινωνικό αποκλεισμό, αλλά πρέπει να σα πω ότι η παρουσία σα ούτω ή άλλω ήταν ενδιαφέρουσα και ιδιαίτερα χρήσιμη. Χρειαζόμαστε τα στατιστικά στοιχεία, χρειαζόμαστε τα στοιχεία από την ε, πραγματικότητα, ώστε να δούμε πώ θα διαμορφωθεί η συζήτηση που έχουμε για την φτώχεια. Σα ευχαριστώ λοιπόν ιδιαίτερω γι' αυτό και θα σα δώσω και πάλι το λόγο για να απαντήσετε όσα περισσότερα ερωτήματα γίνεται. Ευχαριστώ πολύ για την στήριξή σα και για τα πολύ εύστοχα ερωτήματα. Θα προσπαθήσω εν μέρη να απαντήσω και εν μέρη θα δώσω το λόγο στον υπεύθυνο της υπηρεσίας που κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά. Ασχολείται με τα θέματα της φτώχειας. Θα συμπληρώσει τις δικές μου απαντήσεις. Σε πολλές από τις ερωτήσεις. Αναφέρατε σημαντικά προβλήματα συγκρισιμότητας μεταξύ των χωρών και σε διάφορα χρονικά διαστήματα. Μεταξύ των χωρών έχετε απόλυτο δίκιο. Όταν μετρούμε την απουσία πλυντηρίου λόγου χάρη ε, ή για το Λουξεμβούργο και τις κάτω χώρες δεν είναι το ίδιο. Αλλά δυστυχώ είμαστε 27 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν θέλουμε να βρούμε ε, ένα κοινό παρονομαστή για να μετρήσουμε την ηλική στέρηση, θα πρέπει να πάρουμε κάποια συγκεκριμένα αντικείμενα. Αυτό είναι ο μόνο τρόπο να έχουμε συμπεφωνημένου δείκτε μεταξύ των χρηστών των στατιστικών στοιχείων. Βεβαίως, ε, σε γενικές γραμμές ασχολούμαστε με την περαιτέρω βελτίωση της συγκρισιμότητας των δεδομένων. Όμως πρέπει να πω ότι ακόμη και τώρα η συγκρισιμότητα επιτυγχάνεται βάσει των κανονισμών. Οπότε όλες οι χώρες που παράγουν τα δεδομένα βασίζονται σε κοινέ αρχές, σε βασικά και κοινά στοιχεία ε, και ορισμούς από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Οι κανονισμοί λοιπόν που δημοσιεύονται είναι καλής γενικά ποιότητας. Ως προς τους τρεις δείκτες και το πώς περιγράφονται, θέλουμε να έχουμε ένα γενικό προφίλ για να υπάρχει και μια πιστοποίηση ποιότητας για τους δείκτες αυτούς και τη συγκρισιμότητά τους μεταξύ των χωρών. Αυτό είναι μια από τις σημαντικότερες διαστάσεις ε, των ε, σφραγίδων αυτών ε, ποιότητας. Έπειτα αναφέρατε διαφορετικές κατηγορίες του συσχετισμού της στόχιας με άλλες προοπτικές. Λόγω χάρη τη διάσταση της στόχιας από την άποψη της υπαίθρου ή των πόλεων. Ήδη κάποια δεδομένα υπάρχουν για τα θέματα αυτά. Έχουμε πλούσια βάση δεδομένων και τώρα προσπαθούμε να αποσπάσουμε από αυτήν τις χρησιμότερες πληροφορίες μέσω όλων των διαθέσιμων στατιστικών και να τα εκδώσουμε. Ωστόσο, και σε ό,τι αφορά τη διακριτική μεταχείριση λόγω χάρη, πώς να την καταγράψει κανείς εν μέρη ήδη καταγράφεται. Το έδειξα νομίζω αυτό στη διαφάνεια για τους ε, ηλικιωμένους και τα παιδιά. Όμως υπάρχουν και άλλες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού όπως οι μετανάστες, όπως οι ε, άνθρωποι με αναπηρίες. Υπάρχουν και για αυτά κάποιες πληροφορίες και για όσες δεν είναι, το επεξεργαζόμαστε. Λόγω χάρη για τη μετανάστευση έχουμε ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα για το πώ να την, καταγράφουμε. την καταγράφουμε, να την καταπατρώμε για τους μετανάστες συγκεκριμένα και ακόμη και για τη φτώχεια. Ε, για μια από τις ερωτήσεις, ποια είναι η πηγή των πληροφοριών, χρησιμοποιούμε συγκεκριμένες έρευνες του εισοδήματος και των συνθήκων διαβίωσης, όπως λέγονται SILK. Οι έρευνες αυτές είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους των κοινωνικών στατιστικών, που είναι ήδη αρκετά προηγμένες, αλλά εργαζόμαστε για περαιτέρω βελτιώσεις. Ιδίω για να είμαστε και γέρος έτοιμοι. Να μπορούμε να δημοσιεύσουμε μάλιστα τα δεδομένα νωρίτερα. Είναι πολύ δύσκολο το εγχείρημα των κοινωνικών στατιστικών, όμως ήδη έχουμε επιτύχει κάποια πρόοδο, θα κάνουμε ακόμη καλύτερα πράγματα στο μέλλον. Ίσως Ζανίβ να απαντούσε, Λουί μάλλον, ίσως να απαντούσε σε μερικά ζητήματα για τη φτώχεια. Ίσως να μην έχουν καλυφθεί όλα. Thank you. If, if Ευχαριστώ πολύ. Ναι, θα ήθελα να συμπληρώσω αυτά που είπε η Ίνα, λέγοντας ότι τα εργαλεία που ανέφερε, όπως το ε, Silk για παράδειγμα, είναι πρόσφατα, τέσσερα χρόνια υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λίγο κάποιες χρονολογικές σειρές, ε, που προσμετρούν ακριβώς στην εξέλιξη ορισμένων φαινομένων στο χρόνο και μάλιστα από το ένα έτος στο άλλο στις διάφορες χώρες. Το φαινόμενο τώρα της... Ε, του inward poverty. Μιλάμε δηλαδή για τη φτώχεια η οποία ναι μεν αυξάνεται, η οποία ναι μεν βελτιώνεται, αλλά παραμένει στο επίπεδο της φτώχειας. Ε, κάνατε πολλές ερωτήσεις σε σχέση με το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη, τα Υπουργεία θα, θα χρησιμοποιήσουν το τον ε, με δίκτυ... που επιθυμούν για να μπορέσουν ε, να επιτύχουν τους στόχους του... της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το 2020 που είναι η μείωση της φτώχειας. Όμως οι δείκτες που έχουν επιλέξει τα κράτη-μέλη σε εθνικό επίπεδο μπορούν να μετρηθούν και μέσω του εργαλείου SILK. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε τα αποτέλεσμα των εθνικών πολιτικών και μέσω του SILK. Αν πρόκειται δηλαδή για την μακροχρόνια ανεργία, μπορούμε στο πλαίσιο του SILK, ε, στο πλαίσιο του εργαλείου αυτού, να δούμε πώς αυτό το, αυτή η συγκεκριμένη, ε, αυτό το συγκεκριμένο ε, μέτρο ε, βοηθά στην βελτίωση της κατάστασης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, λέει η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ για την παρουσίαση. Θα λάβετε την παρουσίαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υποθέτω. Πολύ, πολύ σύντομα. Είναι πιθανό. Αυτό που είπατε τώρα, να μας το δώσετε και γραπτός να το καταλάβουμε καλύτερα. Μια και δεν είμαστε τόσο εξοικειωμένοι με τις ε, στατιστικές, εκτός από την παρουσία σας, δηλαδή τις συγκεκριμένε παρατηρήσεις. Ναι, όπως είπα, θα είναι στη διάθεσή σας ε, σήμερα το βράδυ. Θα σας στείλουμε με email και θα είναι επισυναπτόμενοι σε ένα email που θα λάβετε. Θα έχετε λοιπόν όλη την παρουσίαση. Το αν θα γράψετε τις απαντήσεις βέβαια είναι δικό σας ε, θέμα. Εγώ δεν θέλω να σας ε, ε, δημιουργήσω μεγαλύτερο φόρτο εργασίας. Τώρα, αύριο ε, προβλέπεται στις 9 η ώρα το πρωί η Φρονσουάζ Καστέξ, ε, κάτι το οποίο τελικά δεν θα λάβει χώρα. Οπότε θα ψηφίσουμε στις 9.30 ώρα το πρωί, 9.30 ακριβώς το πρωί. Αν μπορείτε λοιπόν να, αρχίσετε, να είστε εδώ 9.30 ώρα το πρωί ακριβώς, γιατί θα αρχίσω στις 9.30 ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.